Colleagues, once more, please Αγαπητοί συνάδελφοι, καθίστε παρακαλώ. Είναι μεγάλη χαρά που μπορούμε να ξεκινήσουμε την απογευματινή μας συνεδρία υπό Επιτροπή Ασφάλειας και Άμυνας. Τρία σημεία έχουμε στην ημερήσια διάταξη. Το πρώτο είναι η παρουσίαση μιας μελέτης που έχει δημοσιευθεί για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και συνεργασία με τους ε, νότιους γείτονές μας. Είναι μεγάλη χαρά για μένα που μπορώ να καλωσορίσω τις δύο κυρίες οι οποίες θα πάρουν το λόγο από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Μελετών για την Ασφάλεια, η κυρία Φλωρόνς Γκάουπ, γνωστή σε μας η οποία θα μας παρουσιάσει την μελέτη, καθώς και η κυρία Άννελης Μπάουμπαους. Δεν ξέρω αν Πάουλς, συγγνώμη αν δεν έχω προφέρει σωστά το όνομά σας. Αυτή η παρουσίαση θα ακολουθήσει συζήτηση στις 4 ε, παρα 5 καθότι περιμένουμε τον Sir Julian King, τον Επίτροπο για την Ένωση στον τομέα της ασφάλειας. Θα πάρει το λόγο και θα μας παρουσιάσει τα μέτρα για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και τη συνεργασία με τρίτες χώρες. Θα δώσω το λόγο, δεν ξέρω ποια από τις δύο κυρίες θα πάρει το λόγο πρώτη, η Φλογός Γκάουμπ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε την ευκαιρία να ξαναέρθω. Όπως ξέρετε, σας κάνουμε μια σύντομη περίληψη της μελέτης ε, που έχουμε κάνει και αφορά την καταπολέμηση της ε, τρομοκρατίας ε, και της νότιας γειτονικές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται για μια παρουσίαση η οποία θα έχει λίγο περισσότερα στοιχεία από αυτά που σας έστειλα στις διαφάνειες. Θα ήθελα καταρχήν να παρουσιάσω το φαινόμενο της προοπτικές του. Είναι κάτι που πολλές φορές δεν το κάνουμε, δεν το θέτουμε δηλαδή σε σωστή προοπτική. Ναι, καταρχήν ζούμε σε μια εποχή με μια πρωτοφανή κατάσταση όσον αφορά την τρομοκρατία, με πολλά πλήγματα και θύματα σε σχέση με τις προηγούμενες δεκαετίες, 70 ή το 80 παραδείγματος χάρη. Αυτό είναι όμως η γενικότερη εικόνα. Στην Ευρώπη τα πράγματα είναι διαφορετικά. Αν ε, δείτε τα νούμερα αυτά που έχετε στις, ε, στην οθόνη, οι χώρες που πλήττονται περισσότερο είναι στην Βόρεια Αφρική και στην Μέση Ανατολή. 48% των συνολικών ε, επεισοδίων που αφορούν την τρομοκρατία συμβαίνουν σε αυτές τις δύο περιοχές και το 85% των θυμάτων της τρομοκρατίας είναι μουσουλμάνοι. Κοιτάξτε λοιπόν βεβαίως και την Ευρώπη, ξέρετε τι συνέβη Χτες το βράδυ οι Βρυξέλλες ε, χτυπήθηκαν για άλλη μια φορά. Υπάρχει λοιπόν τρομοκρατία και στην Ευρώπη. Είναι όμως πιο χαμηλά τα επίπεδα σε σχέση με τα επίπεδα της δεκαετίας του 70 και του 80 που ήταν ε, η πολύ σημαντική εποχή όσον αφορά τα χτυπήματα της τρομοκρατίας. Υπάρχουν ε, λοιπόν χτυπήματα που ήταν πολύ πιο σημαντικά τότε σε σχέση με σήμερα στην Ευρώπη. Και αυτό είναι κάτι που δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Θα ήθελα, εδώ βλέπετε τα στατιστικά στοιχεία που αφορούν την Ευρώπη και βλέπετε που είμαστε κάτω δεξιά, υπάρχουν γενικότερες τάσεις, υπάρχει μια αύξηση των τρομοκρατικών χτυπημάτων. Βεβαίως δεν είμαστε στα επίπεδα της δεκαετίας του 70 και του 80 και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το θυμάστε αλλά μην ξεχνάτε ότι όταν μιλάμε για τη Μέση Ανατολή και για τη Βόρεια Αφρική, εκεί βρισκόμαστε στην καρδιά όσον αφορά την, τα χτυπήματα της τρομοκρατίας. Τώρα, για την περιοχή συγκεκριμένα δεν είναι ένα νέο φαινόμενο. Είναι κάτι που γνωρίζουμε που ξεκίνησε ήδη το 1990 στην Αλγερία, στην Αίγυπτο. Τα επίπεδα όμως σήμερα είναι πραγματικά το αποτέλεσμα ή μάλλον η συνέπεια της άνοιξης, της αραβικής άνοιξης. Βλέπουμε λοιπόν να υπάρχει πολιτική πόλωση, ένταση και το φαινόμενο που διαπιστώνουμε σήμερα είναι κατά κάποιο τρόπο η συνέπεια αυτού. Βλέπετε λοιπόν εδώ ότι πρόκειται για το μέτωπο, για την πρώτη γραμμή αυτών των χτυπημάτων. Ποια είναι τα μέτρα ε, για την καταπολέμηση της ε, τρομοκρατίας. Αυτό που θα ήθελα εδώ να αναφέρω είναι τις προτάσεις και τα μέτρα προτείνει η, ο ε, Οργανισμός των Ηνωμένων Καταρχήν, τι είναι αντιτρομοκρατία, αντιτρομοκρατική δράση. Είναι οτιδήποτε μπορεί να προβλέψει ή να καταπολεμήσει μία τρομοκρατική δράση. Βλέπετε εδώ ότι υπάρχει η στρατιωτική αντιμετώπιση, η ασφάλεια, ίσως όχι η στρατιωτική δράση, αλλά ασφάλεια, δηλαδή η εξουδετέρωση τρομοκρατικών ομάδων, τρομοκρατών. Υπάρχει και η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι κάτι που συμβαδίζει με την στρατηγική των Ηνωμένων Εθνών και βασίζεται σε τέσσερις κατευθυντήριες γραμμές, σε τέσσερις πυλώνες. Τι οδηγεί καταρχήν στην τρομοκρατία, δεύτερον πρόληψη και καταπολέμηση, βεβαίως δηλαδή και εμείς έχουμε μια συνιστόσα ασφάλειας, τρίτον δημιουργία δυνατοτήτων υποδομών και δυνατοτήτων για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας και βεβαίως πάντα λαμβάνοντας υπόψη τα ανθρώπινα δικαιώματα, το Συμβασμό των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου. Πάντα θα πρέπει όταν μιλάμε για ασφάλεια, για άμυνα, είναι κάτι που είναι πολύ σημαντικό στα κράτη-μέλη μας. Εμείς όμως στην Ευρώπη έχουμε μια πολύ πιο ε, ολοκληρωμένη προσέγγιση, γιατί αυτή είναι και η λογική μας. Αν κοιτάξετε λοιπόν στις λεπτομέρειες της μελέτης μας, θα διαπιστώσετε ότι Έχουμε όλα αυτά τα μέτρα που παρουσιάζονται με πολλές λεπτομέρειες. Αναλύουμε τους λόγους που οδηγούν στην τρομοκρατία. Όλη η ευρωπαϊκή δέσμευση με τις χώρες της νότιας, της ε, τις νότιες ε, χώρες, Βόρεια Αφρική, αλλά και η Μέση Ανατολή, έχουν σαν σκοπό να διαπιστώσουμε ποιοι είναι αυτοί οι λόγοι που οδηγούν στην τρομοκρατία να έχουμε μια πρόληψη της τρομοκρατίας. Αυτό το κομμάτι λοιπόν δεν το έχουμε αναλύσει με λεπτομέρειες. Αντίθετα, έχουμε αναλύσει τα τέσσερα αυτά συστατικά στοιχεία, στα οποία βασίζεται και η πολιτική των Ηνωμένων Εθνών, βελτίωση του κράτους δικαίου, προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, βελτίωση της περιφερειακής συνεργασίας και βεβαίως πρόληψη και καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Τίποτα από όλα αυτά δεν είναι ένας καθαρά στρατιωτικός στόχος. Το πρώτο που είναι η δημιουργία δυνατοτήτων και υποδομών. Αν κοιτάξετε την ε, έκθεσή μου, Προσπαθώ να κάνω μία περίληψη. Δίνω πολύ συγκεκριμένα παραδείγματα. Μπορώ να σας δώσω κάποια από αυτά, αλλά υπάρχουν πολλά παραδείγματα στη μελέτη. Τι εννοούμε λοιπόν με το πρώτο αυτό ε, στοιχείο, πρώτον καλό και αποτελεσματικό έλεγχο στα σύνορα. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό στην ε, περιοχή, γιατί όπως ξέρετε δεν είναι καθόλου σίγουρα τα σύνορα ούτε στη Βόρεια Αφρική ούτε στην ε, Μέση Ανατολή. Όπως ξέρετε μπορούν να διακινηθούν και όπλα και άτομα. Υπάρχει βεβαίως η γεωγραφική διάσταση. Είναι πολύ δύσκολο να φυλάξει κανείς ένα σύνορο που βρίσκεται στην έρημο αλλά δεν υπάρχουν και οι δυνατότητε στις περιοχές αυτέ, στα κράτη αυτά, έτσι ώστε να είναι ασφαλή τα σύνορα. Βέβαια, σήμερα έχουμε την τεχνολογία. Στην Ιορδανία, παραδείγματο χάρη, με την βοήθεια τη Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει βελτιωθεί η κατάσταση. Όμω μέχρι να ξεκινήσει αυτό το πρόγραμμα συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση υπήρχε ένα κομπιούτερ, ένα ηλεκτρονικό υπολογιστή για τον έλεγχο όλων των συνόρων. Επίση υπάρχει δυνατότητα ελέγχου των ατόμων που φτάνουν με τις αεροπορικές ε, ε, εταιρείες. Υπάρχουν πολλές συνιστώσεις που να βελτιωθούν. Η συνεργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με κάποιες χώρες όπως ο Λίβανος είναι πολύ σημαντική. Όπως ξέρετε ο ρόλος του Λιβάνου με την Συρία σαν γειτονική χώρα είναι εξαιρετικά σημαντικός. Υπάρχουν λοιπόν μέτρα στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, αλλά και στη Βορειοαφρική, στην Τινησία, στην Λιβύη, με τα νέα μέτρα που έχουν ε, υλοποιηθεί για τον έλεγχο των συνόρων. Θα ήθελα επίσης να αναφέρω και στις διάφορες αδυναμίες τις οποίες έχουμε εντοπίσει και η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει τις αρχές της Τινησίας ε, χωρίς να προσπαθούμε πάντα να επιβάλλουμε τις δικές μας λύσεις. Δεύτερο συστατικό στοιχείο, ποινική δράση, δικαιοσύνη, η οποία βεβαίως αποτελεί μέρος της ενίσχυσης του κράτους δικαίου. Στην Τινησία, παραδείγματος χάρη, είναι ένα παράδειγμα Υπερπληθυσμός στις φυλακές 150% στην Τινησία, 300% στο Λίβανο. Τα νούμερα αυτά είναι εντυπωσιακά. Πρόκειται για άτομα που βρίσκονται στη φυλακή, πρόκειται για νέους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται περιμένοντας την δίκη τους. Πρόκειται δηλαδή για προφυλάκηση. Το δικαστικό σύστημα είναι υπερκορεσμένο. Υπάρχουν καθυστερήσεις οι οποίες είναι πολύ δύσκολο να ξεπεραστούν. Προσπαθούμε λοιπόν με τη συνεργασία που έχουμε με τις χώρες αυτές να βελτιώσουμε την κατάσταση. Το ιδανικό βεβαίως ε, θα ήταν να μην βρίσκονται τα άτομα αυτά στις φυλακές αυτές, οι οποίες όπως ξέρετε είναι κέντρα ρίζοσπαστικοποίησης. Δεν θα μπω σε όλες τις ε, πτυχές, τη χρηματοδότηση, την νομοποίηση εσόδων από παράλληλες διαδικασίες, περιφερειακή συνεργασία. Αυτό θα το παρουσιάσει η Άνελης. Νομίζω ότι ξέρετε όλοι ότι και η Βόρεια Αφρική αλλά και η Μέση Ανατολή δεν είναι χώρες και περιοχές που συνεργάζονται εύκολα. Παραδείγματο χάρη, η συνεργασία μεταξύ υπηρεσιών πληροφοριών. Υπάρχει μεγάλη καχυποψία. Προσπαθούμε σαν Ευρωπαϊκή Ένωση να στηρίξουμε τις ε, συνεργασίες μεταξύ υπηρεσιών πληροφοριών με την ε, χρήση της βάσης δεδομένων της Ιντερπολ. Παραδείγματος χάρη για πλαστά και κλεμμένα διαβατήρια 30 εκατομμύρια Το σύστημα της Interpol έχει περίπου 30 εκατομμύρια σημεία ε, εισόδου σε δεδομένα και καταλαβαίνετε ότι οι χώρες αυτές, όπως η Αλγερία, έχουν ε, εδώ και αρκετό καιρό αρχίσει να χρησιμοποιούν τη βάση της Interpol. Είναι όμως μια βάση την οποία χρησιμοποιούν για να ενημερωθούν, για να παίρνουν στοιχεία, αλλά δεν την ενημερώνουν και δεν τη συμπληρώνουν. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να συνεχίσω για τα θέματα της διευκόλυνσης της περιφερειακής συνεργασίας. Ένα πράγμα το οποίο έχει σημασία είναι η προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συνεργαστεί με τις χώρες της περιφέρειας αυτής και να βοηθήσει τις χώρες να συνεργάζονται μεταξύ τους. Αυτό είναι κάτι το καθοριστικό. Ένας από τους τρόπους που το κάνει η Ένωση είναι ένα θα έλεγα δίκτυο παρακολούθησης και ασφαλείας. Υπάρχουν εμπειρογνώμονες σε πόλεις και χώρες της περιοχής οι οποίοι ασχολούνται με τα θέματα της ασφάλειας και κυρίως της τρομοκρατίας και προσπαθούν μέσω του δικτύου αυτού να ανταλλάσσουν πληροφορίες countries they are based in. Um, in this uh, regard, it's also important to mention that um, the EU is trying to involve uh, the Home Affairs Agency. Προσπαθούμε επίσης να συνεργαστούμε με τις εσωτερικές υπηρεσίες παρακολούθησης και γενικά συλλογής πληροφοριών στην περιοχή. Πρέπει να σημειώσουμε εδώ τον ρόλο που παίζει η Interpol και η Europol, οι οποίες εκπαιδεύουν τις δυνάμεις ασφαλείας της περιοχής. Επίσης και το δίκτυο RAM, το οποίο είναι το δίκτυο αντικατασκοπίας. Στα πλαίσια της καταπολέμησης του ακεραιοφρονισμού. Ε, νομίζω λοιπόν ότι το δίκτυο αυτό τώρα ξεκινάει την δράση του μαζί με το Frontex επίσης το οποίο άλλαξε όπως γνωρίζετε η δομή του πρόσφατα και έχει την δυνατότητα να συνεργάζεται με καλύτερο τρόπο με τις τρίτες χώρες. Να επανέλθω στο τέταρτο σημείο. Έχουμε στην έκθεση ένα κεφάλαιο το οποίο ασχολείται ειδικά με το συγκεκριμένο θέμα, ιδιαίτερα με την πρόληψη και την καταπολέμηση ακριβώς των ε, τρομοκρατικών ομάδων. Υπάρχει και σχετική ε, αύξηση, θα έλεγα, των πιστώσεων που διατίθενται προς την κατεύθυνση αυτή σε σχέση με το 2015 υπήρξε αύξηση 150% στον τομέα της αντικατασκοπίας Είναι βέβαια λίγο περίπλοκο να υπογραμμίσει κανείς και να δώσει μια σωστή ιδέα των δραστηριοτήτων οι οποίες διεξάγονται στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας. Είναι κάτι το αρκετά ευρύ ως δίκτυο Υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που παίζουν ρόλο όπως η προώθηση της αμοιβαία συνεργασίας, ε, υπάρχει η προώθηση της κοινωνικής συνοχής, υπάρχουν δράσεις για την βελτίωση της ζωής των νέων το 30% του πληθυσμού των χωρών αυτών είναι από 15 έως 30 ετών και το 50% είναι άνεργοι και αυτό αποτελεί φυσικά μια βάση για τις ε, τζιχαντιστικές ομάδες ε, να ριζοσπαστικοποιήσουν τμήματα του νεανικού αυτού πληθυσμού. και να προσπαθήσουν να επωφεληθούν των δυνατοτήτων και των ευκαιριών. Ο μέσος όρος των ανθρώπων που στρατεύονται στις οργανώσεις αυτές είναι 27 ετών. Είναι λοιπόν ένας από τους στόχους της Ευρωπαϊκής Παρέμβασης στην περιοχή. Ένα άλλο πρόβλημα είναι η πληθυσμιακή σε εισαγωγικά σοφρονιστική κατάσταση Εκεί υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη αντιπαράθεσης με την ριζοσπαστικοποίηση. Ε, στόχος των ε, τρομοκρατικών ενεργειών και ομάδων είναι φυσικά και οι ομάδες των ε, προσφύγων. Υπάρχει ένας πολύ υψηλός αριθμός προσφύγων, ιδιαίτερα στον Λίβανο και την Ιορδανία έχουν, ε, έχουμε να κάνουμε με χώρες που έχουν το υψηλότερο ποσοστό προσφύγων σε όλο τον κόσμο σε σχέση με τον πληθυσμό τους. Και υπάρχουν προβλήματα με τις ένοπλες σειράξεις στην Συρία, στην Ιεμένη. Έχουμε επίσης και τους Παλαιστίνιους, τους νέους Παλαιστίνιους οι οποίοι δεν είναι ενταγμένοι στην κοινωνία της χώρας στην οποία ζουν Προσπαθούμε λοιπόν να παρακολουθήσουμε την κατάσταση η οποία ισχύει στις ε, περιφέρειες αυτές, όχι μόνο τα θέματα όπως αναφέρα ήδη της ισοσπαστικοποίησης, αλλά και άλλους τομείς, όπως ε, η προσπάθεια ένταξης του, των ανθρώπων αυτών, των νέων ανθρώπων ε, στις τοπικές κοινότητες, η συνεργασία ανάμεσα στις κοινότητες που φιλοξενούν τους πρόσφυγες και τους ίδιους τους πρόσφυγες. Μιλάμε για μεγάλες ομάδες ανθρώπων και η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να δημιουργήσει δυνατότητες απασχόλησης για τους πληθυσμούς αυτούς και έτσι να μετριάσει κάπως τις διαφορές που μπορεί να γεννηθούν από την επαφή ανάμεσα στις διαφορετικές κοινωνίες των προσφύγων και των μονίμων κατοίκων. Υπάρχουν και άλλα βέβαια, και άλλοι τομείς που μας απασχολούν, δεν είναι μόνο οι τρεις αυτές ομάδες, αλλά είναι μικρότεροι σε μέγεθος. Ένα τελευταίο σημείο Προσπαθούμε να βελτιώσουμε λοιπόν και τη συνεργασία όπως είπαμε ανάμεσα στις χώρες της περιοχής. Προσπαθούμε να είμαστε συγκεκριμένοι, να καθοδηγήσουμε ε, την συνεργασία των χωρών στην καταπολέμηση της ε, τρομοκρατίας. Έχουμε προχωρήσει σε επαφές με τον Λίβανο και με την Τινησία Προσπαθούμε να το κάνουμε και με τις υπόλοιπες χώρες της Ανατολικής Μεσογείου και ένα από τα συμπεράσματα της έκθεσης, μιας και ο διάλογος προχωρά με ένα αλλά με χαμηλή ταχύτητα, πολλές φορές υπάρχει έλλειψη πολιτικής βούλησης από πλευράς των εταίρων για διάφορους λόγους. Ένας από τους λόγους είναι ότι έχουμε διαφορετική αντίληψη για την αντιτρομοκρατική δράση από ό,τι έχουμε εμείς. Κάποιες από τις χώρες της περιοχής χρησιμοποιούν μια ιδιαίτερο στρατιωτικοποιημένη κατασταλτική αντίληψη για να αντιμετωπίσουν τις ομάδες αυτές Έχουμε και τις ομάδες της κοινωνίας των πολιτών οι οποίες προσπαθούν έτσι ώστε να αναγνωριστούν σαν πλήρης εταίρος στα πλαίσια της καταπολέμησης των ακραίων συμπεριφορών. Νομίζω ότι καλύψαμε τα περισσότερα σημεία της έκθεσης. Σας ευχαριστώ κυρίες και κυρίες. Να ξεκινήσει η συζήτηση. Θα ήθελε η κυρία Λούζινγκ τον λόγο. Όχι, δεν θέλει να πάρει πρώτη το λόγο. Ο κύριος Τάνοκ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα να μάθω σε ποιο βαθμό ε, το trafficking και η σωματεμπορία είναι πηγή εσόδων για τις τρομοκρατικές οργανώσεις. Ξέρουμε τι συμβαίνει στη Λιβύη και για τις περιοχές τις οποίες ελέγχει η Λιβική Ίσης. Και ένα άλλο θέμα το οποίο με ανησυχεί ιδιαίτερα, μια και από το Ηνωμένο Βασίλειο, είναι το ποιες θα είναι οι συνέπειες του Brexit. Δεν ξέρω αν έχει δοθεί προσοχή ε, στο πώς η χώρα μου θα συμμετέχει σε όλες τις πρωτοβουλίες τις οποίες αναφέρατε. Στην έκθεσή μου είχα απευθύνει την έκκληση το Ηνωμένο Βασίλειο να παραμείνει κομμάτι αναπόσπαστο του πλαισίου μέσα στο οποίο αντιμετωπίζουμε θέματα τέτοιου είδους και απειλές τέτοιου είδους. σαν παράδειγμα PNR, ε, Eurojust, ε, Europol, ε, Eurodact, δεν ξέρω ποια θα είναι η συνέχιση της συνεργασίας μετά το Brexit. Λόγω του σταδιακού χαρακτήρα των διαπραγματεύσεων και λόγω των θεμάτων ασφαλείας τα οποία θα τεθούν προς συζήτηση στην δεύτερη φάση, απαιτείται να υπάρξει σημαντική πρόοδος στην πρώτη φάση ανάμεσα στους εταίρους και τίποτα δεν θα έχει συμφωνηθεί αν δεν συμφωνηθούν όλα. Και υπάρχει συνεπώς ο κίνδυνος ε, μιας, ενός καινού ασφαλείας. Θα ήθελα αν δεν υπάρξει μια αμοιβαία μορφή κατανόηση, μια κοινή κατανόηση του Brexit να αναγνωρίσουμε τους κινδύνους που δημιουργούνται για την ευρωπαϊκή πλευρά ε, και για το Ηνωμένο Βασίλειο και το λέω αυτό και ως εκπρόσωπος των φιλοευρωπαίων του Συντηρητικού Κόμματος. Ο κύριος Μποστινάρου έχει το λόγο. Τώρα για τις δυνατότητες οικοδόμησης κρατικών θεσμών. Ποιες είναι οι προκλήσεις τις οποίες έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Υπάρχουν ορισμένες ασθενείς χώρες ή χώρες υπό αποτυχία ή θα έλεγα καλύτερα σε διαδικασία αποσύνθεσης. Πώς είναι σε θέση να συνεργαστούν με δυνατότητες αντιτρομοκρατικέ ε, και με συνεργασίες ε, και πώς μπορούμε να τις βοηθήσουμε τις χώρες αυτές. Και δεύτερον, τι προσοχή δίδουμε εμείς έτσι ώστε να αποτρέψουμε τις υπηρεσίες αυτές να καταστούν αυστηρά κατασταλτικά μέσα εξυπηρέτησης των πολιτικών οδηγιών των ηγετών τους. Ένα δεύτερο θέμα. Θα ήθελα και εγώ να θέσω την ερώτησή μου, αν δεν σας πειράζει. Κοιτάξτε, να περιοριστώ σε μία ακόμα ερώτηση. Στα πλαίσια ε, της καταπολέμησης της ε, τρομοκρατίας ε, αυτές, σε αυτές τις χώρες. Τι ρόλο μπορεί να παίξουν οι, ο, ο κλήρος των, μουσουλμάνων και της θρησκευτική εξουσίας έτσι ώστε να υπάρξει μια μεταρρύθμιση της εικόνας του Ισλάμ προς τα έξω και σαν παράδειγμα οι θέσεις ε, του Προέδρου της Αιγύπτου και η έκκλησή του για τον εξυγχρονισμό της ψυχής του Ισλάμ όπως είπε. Και δεύτερον ποιος είναι ο ρόλος των αυτοανακηρυγμένων ημάμιδων ε, στον διαδικασία ριζοσπαστικοποίησης και στράτευσης. Είναι σημεία τα οποία ενδιαφέρουν τις χώρες αυτές αλλά ενδιαφέρουν και εμάς. Έχουμε και εμείς πρόβλημα. Ο κύριος Φρόιντ. Χαιρόμαστε που σας ξαναβλέπουμε, Φλόρενς. Δύο ερωτήσεις. Κατά κάποιο τρόπο επί της ακμής των όσων συζητήσατε. Πρώτα, η ιδέα που συζητείτε κάποιο διάστημα τώρα, μετά από τα 70 χρόνια του σχεδίου Μάρσαλ εδώ στην Ευρώπη. Μια ασαφής μεν έννοια, μια ιδέα να γίνει κάτι παρόμοιο για χάρη της Αφρικής, που ίσως θα προλάβαινε όλα αυτά που λέτε. Τι πιθανότητες επιτυχίες δίνατε σε κάτι τέτοιο και τα χρήματα, εφόσον αυτό είναι το ουσιώδες μέρος του σχεδίου Marshall εντό εισαγωγικών, αλλαγής μπορεί να επιφέρει το χρήμα. Δεύτερη ερώτηση, ελπίζω να μην την ξέχασα. Είναι άλλο θέμα. Ιδιαίτερα ενδιαφέρον στην Αυστρία τώρα, συζητείται πολύ έντονα, η ιδέα ότι τα όσα κάνατε την οδό των Δυτικών Βαλκανίων που την κλείσατε και τώρα το ερώτημα είναι αν όντω έχει κλείσει ή εάν η Τουρκία δεν αποστέλει πλέον μετανάστες μέσα από την οδό αυτό προς την Ευρώπη. Και αυτό οδηγεί στο ότι τελικώ την ε, οδό αυτή την παίρνουν λιγότεροι μετανάστες. Αλλά πώς αυτό μπορεί να εφαρμοστεί και, ε, και στην Μεσόγειο, στην οδό της Μεσογείου. Αντιλαμβάνομαι ότι δεν είναι αποκλειστικά τη αρμοδιότητά σα, αλλά είστε εμπειρογνώμων επιγενικών θεμάτων άλλωστε και μήπω έχετε κάποια ιδέα. Πώ ε, δηλαδή θα μπορούσε να διαχειριστεί κανεί κάτι τέτοιο και αν είναι καν διαχειρίσιμο. Η κυρία Φωτίγκα, ε, κάπως όπως και ο κύριος ε, Φρόιντ, θα ήθελα να πω και εγώ ότι βρισκόμαστε σε μια συζήτηση για το θέμα αυτό. Πώς περιγράφετε εσείς αυτό το modus operandi μεταξύ ορισμένων χωρών της νότιας γειτονίας, τις οποίες περιλαμβάνονται και κάποιες χώρες διεύρυνσης στη συνεργασία με την Τουρκία όσον αφορά την ανακοπή των μεταναστευτικών ρευμάτων. Πώς μπορείτε να περιγράψετε την ε, συνεργασία και για τον εντοπισμό τρομοκρατών στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε τι επίπεδο κινείται η συνεργασία αυτή. Αυτό νομίζω ότι, μάλλον νομίζω ότι η συνεργασία αυτή είναι ομαλή, παρά τις κάποιες εντάσεις και συνεχίζεται η εμπλοκή αυτή. Πώς μπορείτε να περιγράψετε τη συνεργασία με το Μαρόκο, για παράδειγμα. Σε ό,τι αφορά την Τινησία, ακούσαμε από τα μέσα ενημέρωσης και στη διερεύνηση των τρομοκρατικών επιθέσεων σε διάφορες χώρες της Ένωσης. Μάθαμε ότι συνεργάζονται ή τουλάχιστον αντιλαμβάνομαι ότι είναι διατεθειμένες οι αρχές τους να συνεργαστούν. Πληροφορίες τώρα και παρατηρήσεις που κάνατε σχετικά με τον Λίβανο. Υπάρχει κάποια γραμμή συνεργασίας με την έννοια όχι μόνο να προσφέρουμε σταθερότητα και ασφάλεια, να μπορούμε και να διδαχτούμε κιόλας. Θα ήθελα να ακούσω την άποψή σας Επίσης σχετικά με τη συνεργασία με το Ισραήλ για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Ποιες διαφορές εντοπίζεται στις προσεγγίσεις, πού βρίσκονται ομοιότητες και πού ενδεχομένως ανοίγεται ένα πεδίο συνεργασίας. Ο κ. Νάρτου y coincido plenamente con la pregunta de un compañero. Ήθελα να απαντήσω. Τριπλή ερώτηση. Η δημιουργία αυτών των δημιουργείται στη Μεσκίτα Μοχάμετ στην Καζαμπλάνκα, αυτή η νέα σειρά ημάμιδων, που είναι μια πλατφόρμα θα έλεγα μηχανισμοί όπως είπα ακραίων ε, και υπάρχουν αυτόνομοι μεντρεστέδες οι οποίοι παράγουν οι μάμιδες οι οποίες μαζεύουν τα παιδιά που δεν έχουν μέλλον, τα παιδιά που έχουν εγκαταληφθεί από τις οικογένειές τους και προσπαθούν να ξεφύγουν από ένα διεφθαρμένο περιβάλλον και να βρουν κάποιο μέλλον μέσα ακριβώς σε αυτήν την πρωτόγονη ερμηνεία του Ισλάμ. Δεύτερον, ποια είναι η άποψή σας για τις δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Λιβύη. Ο συνέτερός μας είναι ο Φαράς, τον οποίο κανένας δεν αναγνωρίζει εκτός από τους Γάλλους, τους Ισπανούς, τους Πολωνούς και τους Αμερικανούς. Αλλά δεν τους αναγνωρίζουν οι ίδιοι οι Λίβοι. Οπότε πώς ακριβώς συνεργαζόμαστε με αυτούς. και η βοήθεια την οποία δίδουμε στις περιοχές αυτές δεν έφτασε ποτέ ούτε στην Τρίπολη, ούτε στη Βεγγάζη, ούτε στο Πομπούκ. Και τέλος, τι γίνεται με την α, ακτοφυλακή την οποία χρηματοδότησε η Ευρώπη σε αυτά τα λιμάνια, ε, λιμάνια τα οποία πολλοί ελέγχονται από το οργανωμένο έγκλημα. Πρόκειται ε, για αστυνομικές υποτίθεται δυνάμεις ε, οι οποίες όμως εξυπηρετούν ουσιαστικά τα συμφέροντα του ε, παράνομου χώρου του, των εγκληματικών δραστηριοτήτων συνεργάζονται αυτά τα στοιχεία της ακτοφυλακής με, τις, με τους εκπροσώπους του οργανωμένου εγκλήματος μόνο και μόνο γιατί το οργανωμένο έγκλημα επιτρέπει στα παιδιά τους και την οικογένειά τους να μείνει ζωντανή. Υπάρχουν έξι ένοπλες ε, δυνάμεις στην χώρα αυτή ε, που στην ουσία είναι κάτι το οποίο δεν ε, μας δίνει την δυνατότητα αποκατάστασης σχέσεων μαζί τους. Okay. Η πρόεδρος Φωτίγκα. Ε, εσείς κυρία Κάουπ, σας ευχαριστώ για τις ενδιαφέρουσες ερωτήσεις. Θα προσπαθήσω να τις απαντήσω με τη σειρά που τις υποβάλλατε. Για τη σωματεμπορία και για την χρηματική διάσταση θα σας τα πει συναδελφός μου. Ό, όταν αποφασίστηκε το Brexit ήμουν πεπισμένη ότι η Βρετανία θα παραμείνει σημαντικό μέρος της αμυντικής αρχιτεκτονικής ή πάντως του αμυντικού χώρου στην Ευρώπη. Με τον ίδιο τρόπο που κατά κάποιο τρόπο είναι και οι Ηνωμένε Πολιτείε μέρος του Ευρωπαϊκού Αμυντικού Χώρου. Βλέπει Ευρωπόλ, ε, ανταλλαγή δεδομένων ε, αλλοδαπών μαχητών και άλλες ιστορίες. Ε, εν τέλει, βέβαια βρίσκεται στα χέρια του κυρίου Μπαρνιέ και τον συναυτό το πώς θα διαμορφωθεί τελικά αυτή η σχέση. Είναι αδιαμφισβήτητο και παριμήν και παριμήν με ύπτα και ύψιλον ότι θέλουμε να συνεχίσει η ανταλλαγή πληροφοριών. Ξαναλέω ότι είναι αδιαμφισβήτητο και είναι και σημαντικό και ουσιώδες. Λιβύη. Πώς ξανά ε, στα πόδια της κανείς μια χώρα, ένα κράτος το οποίο έχει ε, ε, καταστραφεί. Αυτό είναι πολύ δύσκολο. Εάν κοιτάξετε την περίπτωση του Ιράκ ή και τη Λιβύη, αν δεν έχετε θεσμούς που να μπορείτε να τους χρησιμοποιήσετε για να οικοδομήσετε από αυτόν, θα χρειαστεί πάρα πολλή χρόνο, θα είναι πολύ ασταθές το κράτος αυτό μέχρι ότου επιτύχει τον στόχο και βεβαίως θα είναι εξαιρετικά δαπανηρό. Ε, μιλώ για το Ιράκ διότι αρχικά το σχέδιο ήταν να ξαναρχίσει ο Ιρακινός στρατός από το μηδέν μετά από το Σατάμ Χουσέιν. Μετά όμως η έλλειψη ασφάλειας οδήγησε στο συμπέρασμα ότι αυτό δεν ήταν δυνατό. Ξανάφεραν λοιπόν στο στράτευμα πολλούς Ιρακινούς αξιωματικούς και στη Λιβύη τα απομεινάρια του Λιβικού στρατού που ήταν σε πολύ χειρότερη κατάσταση και από τον Ιρακινό στρατό πριν από το 2011 τώρα μάχονται στον πρώτο χάφτα. Αλλά είναι όμως ηλικιωμένοι άνθρωποι είναι συνταγματάρχες και δεν έχουν και μεγάλη όρεξη να ασχοληθούν με τους παρακάτω βαθμούς. Είναι λοιπόν ένα δύσκολο ένιγμα. Η δύσκολη αλήθεια είναι ότι ή περιμένει κανείς μέχρι ότου ισορροπήσουν τα πράγματα, μέχρι ότου κουραστούν να μάχονται με τους δε δηλαδή, είτε στέλνεται μια ηρωνοποιό δύναμη και τους επιβάλλεται την ειρήνη. Πολύ δύσκολη υπόθεση και πολύ δαπανηρή. Και ούτε βλέπω κανένα να έχει όρεξη να το κάνει αυτό τώρα. Το άλλο ε, σημαντικό ε, σε σχέση και με την, τον πολιτικό πολιτισμό της Λιβύης δεν είναι ίσως ακριβώς αποτυχημένο κράτος η Λιβύη, διότι αυτό που βλέπετε στη Λιβύη σήμερα είναι, ε, εξακολουθούν, να υπάρχουν της τζαμαχηρία, κάτι που είχε επινοήσει ο Καντάφη και εξακολουθούν και λειτουργούν. Αυτά τα βασικά συμβούλια 450 στη, σε ολόκληρη τη χώρα ξεχνούν και λειτουργούν και παίρνουν αποφάσεις και διαχειρίζονται θέματα όπως η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, νερού κτλ. Εκεί που δεν λειτουργούν είναι στις περιοχές εκείνες όπου είναι και ο ίδιος ο Καντάφη. Δεν άντεξαν τα συστήματα αυτά, ιδίως στους χώρους της ασφάλειας, άμυνας και εξωτερική πολιτικής. Διεύρωσε το κράτος αυτό λοιπόν, ο Καντάφη σε αυτούς τους κέρδους τομείς. Και εκεί παλεύει η Λιβύη και δεν τα καταφέρνει τώρα και θα χρειαστεί κάτι περισσότερο από μια ειρηνευτική δύναμη για να ξαναδημιουργήσει αυτό το πολιτικό πολιτισμό. Και στο μεταξύ βέβαια υπάρχει το πρόβλημα όπως είπατε και εσείς. Για το ισπανικό ερώτημα, αλλά βέβαια για την ε, λιβική ακτοφυλακή, πήγα να πω ισπανική ακτοφυλακή, έχετε δίκιο. Παίζουν, μάλλον τα καλά νέα είναι ότι πολλοί προερχόνται από το παλαιό καθεστώς και επομένω έχουν κάποια γνώση για το πώς γίνονται τα πράγματα. Αλλά προχωρούν σε συμπεγνία με τους ε, λαθροδιακινητές. Ε, μπαίνουν ε, μέσα στην υπόθεση αυτή και στις συμφωνίες αυτές και κάποια δίκτυα φυλών της χώρα αυτής. Ακόμα και αν έχετε ένα τέλειο σχέδιο οργανογράμματος για την ακτοφυλακή και προσπαθεί να το επιβάλλεται. Για παράδειγμα το γεγονός ότι για μας για μας ο έλεγχος των συνόρων είναι καθήκον της αστυνομίας. Για τους Λίβιους ο έλεγχος των συνόρων είναι καθήκον του στρατού. Υπάρχουν λοιπόν ορισμένα πράγματα που ε, για εμά του Ευρωπαίου είναι διαφορετικά. Έτσι είμαστε εμεί, έτσι κάνουμε τη δουλειά μας, αλλά η κατάσταση επιτόπου είναι πάρα, πάρα πολύ διαφορετική από αυτά που γνωρίζουμε εμεί εδώ. Το ερώτημα Ε, το γεγονός λοιπόν ότι χρησιμοποιούν τι χρηματοδοτήσει μας για δικές τους δράσεις και όταν υπάρχει από την άλλη μεριά άρνηση όπως στην Αίγυπτο δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Και είναι μεγάλη ανησυχία η Αίγυπτος όχι μόνο λόγω των φυλακών, λόγω των μαζικών δικών και καταδικών. Η μεγαλύτερη ανησυχία είναι ότι αυτά όλα δεν αποδίδουν καν. Και αν θα ήθελε κανεί να τα δει κοινικά, θα μπορούσε να πει κανείς «Α, είναι βέβαια ε, η δράση τους κατασταλτική, αλλά αποδίδει». Αλλά δεν αποδίδει, είναι δικτάτορες και χειροτερεύει και το πρόβλημα. Ως Ευρωπαίοι λοιπόν ανησυχούμε για το θέμα αυτό, το θέτουμε, προσπαθούμε να το θέσουμε και σε όλα τα επίπεδα και ενώπιον των Αιγυπτίων και ενώπιον άλλων για να τους το υπενθυμίσουμε, αλλά εν τέλει η Αίγυπτος είναι κυρίαρχο κράτος και έχουν το προνόμιο της κυριαρχίας. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε περισσότερο. Για το σχέδιο Μάρσαλ Κύριε Φρόιντ, ευχαρίστως δέχομαι αυτό που είπατε. Σχέδιο Μάρσαλ για την περιοχή αυτή. Και ο Ιταλός Πρωθυπουργός στο G8 είχε προτείνει την ιδέα, αλλά μέχρι εκεί έφτασε η ιδέα αυτή. Και ο βασικός λόγος είναι ότι το σχέδιο Μάρσαλ είχε και μια διάσταση ασφαλείας και ήταν σαφές ότι τα χρήματα θα επιστρέψουν. Κράτη και επιχειρήσεις δεν θέλουν να επενδύσουν στη Μέση Ανατολή διότι δεν θεωρούν ότι θα ξαναπάρουν ποτέ πίσω τα λεφτά τους. Προτιμούν να επενδύουν, για παράδειγμα, στην πετρελοβιομηχανία, όπου γνωρίζουν ότι θα αποδώσουν τα κεφάλαια αυτά. Αυτό που έχει κάνει η Ευρώπη τα τελευταία χρόνια είναι ότι έχει φτιάξει ένα ευρωπαϊκό, νομίζω, επενδυτικό σχέδιο, όπου οι επενδυτές καλύπτονται. Υπάρχει δηλαδή μια κάλυψη για τις εταιρείες που επιθυμούν να επενδύσουν. Foreign direct investment δηλαδή είναι αυτό το οποίο θα μπορέσει να οδηγήσει σε δημιουργία απασχόλησης και καινοτομίας. Και προ τα εκεί θα πρέπει να κατευθυνθεί. Το σχέδιο αυτό συζητήθηκε ήδη τον Νοέμβρη και νομίζω θα ήταν πραγματικά καλή ιδέα. Για την οδό των Δυτικών Βαλκανίων και μετά να περάσω αν το μικρόφωνο στη συναδελφό μου, η μόνη χώρα επί του παρόντος που βρίσκεται στο επόμενο σταυροδρόμι των μιζώνων μεταναστευτικών ροών είναι η Αίγυπτος. Οι Αιγύπτιοι καλά τα καταφέρουν για την ώρα στον έλεγχο των σημείων εξόδου. Είναι πολύ μικρότερη η λαθροδιακίνηση από την Αίγυπτο, από την, από Λιβύη. Αυτό που μας ανησυχεί όμως είναι ότι εάν έχουμε άλλη μια μεγάλη κλίμακα εξέγερση όπως είχαμε το 2010-2011, δεν θα αντέξουν οι ελέγχοι αυτοί και θα αρχίσουν οι ροές μέσω της Αιγύπτου, διότι τα δίκτυα υπάρχουν ήδη τόπου και είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να μας ανησυχεί και γι' αυτό η συνέχιση του διαλόγου με τους Αιγυπτίους ανεξαρτήτως του πώς διαμορφώνεται η κατάσταση είναι πολύ σημαντικό. Τέλος. Για την ηχνηλάτηση έλλειψη συνεργασίας μεταξύ των χωρών της περιοχής αυτής για την ανταλλαγή πληροφοριών. Όλες οι χώρες έχουν πρόβλημα με τους γείτονές τους και δεν ανταλλάσσουν πληροφορίες. Θέλουν κάποιος, ε, κάποιον να απελάσουν. Ήδη από το 1996 ε, Αλγερία, Μαρόκο έχουν κλειστά σύνορα. Ε, το ίδιο άλλες χώρες. Ιράκ και Σαουδική Αραβία. Κλειστά τα σύνορα του μεταξύ του εν τέλει. Πολλές από τι τράπεζε δεδομένων δεν είναι διασυνδεδεμένε των χωρών αυτών και πολλέ από τι διελεύσει των σύνορων δεν έχουν ηλεκτρονικού υπολογιστέ. Αν είστε λοιπόν λάθροδιακινητής ή λαπαράνομος ή οτιδήποτε, μπορείτε να περάσετε. και είναι και δύσκολο να εντοπιστούν και οι επιστρέφοντες άλλο μαχητές. Τελειώνω με το Ισραήλ. Έχουμε συνεργασία σε έναν βαθμό με το Ισραήλ, αλλά όπως ξέρετε είναι κάπως διαφορετική η ερμηνεία. Αν θυμηθείτε και τα τέσσερα σημεία που σας εξήγησα, και η τρομοκρατία στο Ισραήλ έχει διαφορετική απόχρωση από αυτήν που αντιμετωπίζουμε εμείς εδώ ή άλλες χώρες της περιοχής αυτής. Διότι ως τώρα το Ισλαμικό κράτος δεν έχει καταφέρει να στρατολογήσει Παλαιστινίους. Και αυτό διότι η Παλαιστινιακή τρομοκρατία κινείται από εθνικά συναισθήματα ανεξαρτησίας κλπ. Για τους Ισραηλινούς λοιπόν, λοιπόν είναι διαφορετικό το πρόβλημα και είναι βέβαια πάρα πολύ έντονη η ε, ε, διάσταση της αποτροπής με πολύ βαριά καταστολή, ε, ποινές φυλάκισης, καταστροφές οικειών κτλ. Έτσι λοιπόν ερμηνεύουμε η πλευρά των Ισραηλών και εμείς με διαφορετικό τρόπο την αντιτρομοκρατία. Η πρώτη ερώτηση που θα απαντήσω είναι αυτή που αφορά την τρία διακίνηση μεταναστών. Βεβαίως αυτό έχει άμεση σχέση με την τρομοκρατία, ιδιαίτερα στις περιοχές που εξετάζουμε σήμερα. Και βεβαίως όσον αφορά τα προηγούμενα μέτρα που έχουν ληφθεί, όσον αφορά την ειδική ομάδα για τη χρηματοδότηση η οποία συστάθηκε αμέσως μετά την επίθεση την 11η Σεπτεμβρίου και όλη αυτή η δράση για την πρόληψη της χρηματοδότησης είτε από ιδιώτες είτε από κρατικές αρχές. Όπως ε, ξέρετε είναι σε θέση οι ομάδες αυτές ε, να βρουν χρηματοδότηση και κυρίως αυτό γίνεται μέσω εγκληματικών ε, δραστηριοτήτων κάθε είδους όπως ξέρετε διάφορα προϊόντα, ναρκωτικές ουσίες, καπνός, προϊόντα καπνού, όπλα και γνωρίζουμε ότι αυτού του είδους οι εγκληματικές δραστηριότητες χρηματοδοτούν την τρομοκρατία. Είναι επίσης ε, ένα σχέδιο το οποίο κυρίως θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με συνεργασία με τρίτες χώρες, ιδιαίτερα προσπαθώντας να διακόψουμε και να σταματήσουμε αυτή τη χρηματοδότηση της ε, τρομοκρατικής δράσης. Αυτή είναι μία από τις προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε, ιδιαίτερα όσον αφορά γενικότερα τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Και εδώ, όπως είπε και η Φλογός, Ακριβώς επειδή δεν υπάρχει πραγματική ανταλλαγή πληροφοριών, ε, η δράση μας είναι περιορισμένη. Στην ε, περιοχή, παρόλα αυτά, υπάρχουν διαφορετικές νομοθεσίες ε, που αφορούν την καταπολέμηση της τρομοκρατίας από τη μια χώρα στην άλλη και υπάρχουν, θα έλεγα, πολλά κενά αδύναμα σημεία Πολλές φορές οι αρχές της μιας χώρας δεν γνωρίζουν τις διαφορές της νομοθεσίας μιας γειτονικής τους χώρας, δεν ξέρουν πώς να υποβάλουν, παραδείγματο χάρη ένα αίτημα δικαστικής συνδρομής, πολύ απλά και πρακτικά θέματα τα οποία δεν έχουν καν σχέση με τη γενικότερη πολιτική του ενός ή του άλλου κράτους, που δεν είναι σε θέση να τα διεκπαιρεώσουν χρειάζεται σε κάθε περίπτωση αυτή η νομική συνεργασία για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε ε, με αποτελεσματικό τρόπο την χρηματοδότηση της ε, τρομοκρατίας. Άλλες προκλήσεις υπάρχουν χώρες που σαφώς και λειτουργούν, η οικονομία τους λειτουργεί με τις ε, συναλλαγές χρησιμοποιώντας ε, ρευστότητα και βλέπουμε ότι το ρευστό χρήμα είναι πολύ πιο εύκολο να χρησιμοποιηθεί σε τέτοιου είδους εγκληματικές δραστηριότητες αλλά και για την νομιμοποίηση παράνομων ε, πόρων. Και αυτό είναι ένα ε, ευρύτατο φαινόμενο στην περιοχή. Μιλήσατε επίσης και για τους αυτοδιοριζόμενους ε, ημάμιδες και το ρόλο τους στην ριζοσπαστικοποίηση. Δεν ξέρω αν ε, είναι σωστό να δούμε την ε, ριζοσπαστικοποίηση από αυτή την οπτική γωνία. Τα τελευταία δέκα χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε προσπαθήσει να δούμε τι ρόλο παίζουν αυτοί οι εκπρόσωποι της θρησκείας αυτής στην ριζοσπαστικοποίηση νέων, ποιος είναι ο ρόλος των πιο μετριοπαθών ε, μουσουλμάνων, το θέμα των ε, στερεοτύπων και δεν είναι, αν θέλετε, σήμερα σαφές το κατά πόσο αυτοί οι συγκεκριμένοι ε, εκπρόσωποι της μουσουλμανικής θρησκείας παίζουν έναν καθοριστικό ρόλο στην ε, ριζοσπαστικοποίηση. Σίγουρα ε, ο ρόλος της θρησκείας είναι σημαντικός, αλλά δεν πιστεύω ότι είναι ο πιο σημαντικός. Παραδείγματος χάρη, πολλοί από αυτούς οι οποίοι επέστρεψαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση αφού προηγουμένως είχαν ε, πάει στην Συρία και πολέμησαν με τους μαχητές του Ντάες. Οι περισσότεροι από αυτούς δεν είχαν μεγάλη επαφή με τη θρησκεία. Ο ρόλος λοιπόν των ε, ημάμιδων στην ε, ριζοσπαστικοποίηση ή στη στράτευση είναι περιορισμένος κατά την άποψή μας. και θεωρούμε ότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και το διαδίκτυο δίνουν σήμερα άλλες δυνατότητες ε, στους ε, νέους που θέλουν να προσχωρήσουν για να ριζοσπαστικοποιηθούν από μόνοι τους. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Νομίζω ότι έχουμε ολοκληρώσει. Ο κύριος Τάνοκ όμως θέλει να κάνει άλλη μια ερώτηση. Πολύ σύντομα, κυρία Πρόεδρε. Αυτό που άκουσα με άφιασε κατά κάποιο τρόπο, ότι δεν υπάρχει δηλαδή συνεργασία των υπηρεσιών πληροφοριών μεταξύ των κρατών της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής. Εδώ όσον αφορά την αραβική τον Αραβικό Σύνδεσμο και άλλες διεθνούς οργανισμούς πώς θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε αυτήν την ε, έλλειψη συνεργασίας. Ξέρουμε ότι υπάρχει βεβαίως και μια ιστορική εξήγηση. Ε, οι πολύ κακές σχέσεις που έχουν οι αραβικές χώρες μεταξύ τους και μεταξύ του Ισραήλ και των γειτονικών χωρών. Σαφώς ε, όμως μπορεί να βελτιωθεί η κατάσταση. Εγώ ξέρω ότι και στις δικές μας χώρες η ανταλλαγή πληροφοριών είναι δύσκολη. Παραδείγματος χάρη μεταξύ Γαλλίας και Βελγίου όπως είδατε, υπήρξαν προβλήματα με την ανταλλαγή πληροφοριών και μετά την επίθεση στον Πατακλάν. Σίγουρα θα πρέπει εδώ να ασκηθεί πίεση, όπως είπα, από τους διεθνείς οργανισμούς, τον Αραβικό Σύνδεσμο, τους οργανισμούς αυτούς, στους οποίους συμμετέχουν οι χώρες αυτές για να υπάρξει πραγματική ανταλλαγή πληροφοριών. Είναι προφανές ότι δεν μπορεί κανείς να υποδομήσει στο τίποτα. Στην περίπτωση της Λιβύης, όπως είπατε, ε, ο Λιβικός στρατός ε, είναι παλαιοί πολεμιστές, ε, αλλά εγώ μπορώ να σας πω γιατί έχω, τους έχω δει από κοντά. Μπορώ να πω ότι μάχονται σαν νέοι, δεν είναι βέβαια εκλεκτά στρατεύματα, αλλά πάντως μπορούν να δώσουν μάχες ιδιαίτερα σε σχέση με την δυνατότητα που έχουν να ανακαταλάβουν τις περιοχές τις οποίες ελέγχει το χαλιφάτο. Ξέρετε πόσες φορές έχουν αντισταθεί στην κατάληψη του, ε, με του το στο οποίο είναι εγκατεστημένο στο Ελαράς. Θα ήθελα λοιπόν να μάθω αν πράγματι ακούγοντας και όλα αυτά τα οποία είπατε για τους ημάμιδες και την ριζοσπαστικοποίηση του Ισλάμ. Ένα θέμα είναι η Ευρώπη, ένα άλλο είναι η Αφρική. Υπάρχουν οι αυτόνομοι ε, μεντρεσέδες των αναλφάβητων, αμόρφωτων ημάμιδων. Παίζουν δυστυχώς ε, παίζουν σημαντικότατο ρόλο στην ε, ζώνη κάτω από το ΣΑΕΛ αν δεν δημιουργηθούν νέοι ημάμιδες, αν δεν ευνοηθεί η δημιουργία νέων ημάμιδων, τότε ε, ο ριζοσπαστικός χαρακτήρας του Αλισλάμ και του Μπόκο Χαράμ θα κυριαρχήσει στην περιοχή από τον Ήγηρα μέχρι το Τσάδα. Και ο τζιχαντισμός ε, δυστυχώς θα γίνει ένα καθολικό φαινόμενο και όχι απλά ευρωκεντρικό και στη συγκεκριμένη περίπτωση όλος αφρικανικό. Πρέπει λοιπόν να δούμε ποιος είναι ο ρόλος των ανεξάρτητων αυτών αυτών ημάμιδων στην εκπαίδευση και την προετοιμασία άλλων. Ο Επίτροπος Κίνγκ είναι ήδη εδώ για το επόμενο θέμα. Νομίζω ότι μπορούμε να το θέσουμε εκ νέου το θέμα. Μπορείτε να παραμείνετε αν θέλετε, όχι πρέπει να φύγετε. Λοιπόν, ε, ο Επίτροπος θα μας επιτρέψει μια πολύ σύντομη απάντηση. Συγγνώμη. Πρέπει να φύγουμε σε μια άλλη διάσκεψη όπου έχουμε ένα δεκάλεπτο μόνο στη διάθεσή μας. Αυτό το οποίο έχει σημασία ε, ότι αντίθετα με τον Ιουδαϊσμό σαν παράδειγμα, ε, το Ισλάμ δεν έχει μια επίσημη διαδικασία Εκπαίδευση και κατάρτιση των ημάμιδων. Το ημάμ, η ίδια λέξη έρχεται από τη λέξη αλμάμα που σημαίνει το να είσαι μπροστά, το να είσαι πρωτοπόρος. Συνεπώς λοιπόν μπορείς να ορίσεις τον εαυτό σου ως ημάμι και αν υπάρχει μια ομάδα η οποία λέει ότι λες την αλήθεια τότε καθιερώνεσαι ακόμα και αν λες σαχλαμάρες. Έχουμε ένα πρόβλημα διαγενειακό όπως είπε η Άνελης ε, κάποιοι παλαιοί ημάμιδες πλέον δεν έχουν την δύναμη την οποία έχουν στην διάθεσή τους τώρα οι ριζοσπαστικοποιημένοι ημάμιδες. Για τη Λιβύη συμφωνώ μαζί σας αλλά δεν μπορώ τώρα να περάσω σε λεπτομέρειες. Η σημερινή παρουσίαση έχει σχέση με την συνεργασία για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Γενικότερα για την τρομοκρατία μπορούμε να τα πούμε σε μια άλλη ευκαιρία. Σας ευχαριστώ. Περνάμε τώρα στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Στην ουσία θα υπάρξει μια συνέχεια, αν θέλετε, του ιδίου ε, θέματος της ίδιας συζήτησης. <laughs> interesting. We going to Πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Θα συνεχίσουμε κατά κάποιο τρόπο τη συζήτηση. Το θέμα τώρα είναι λίγο ευρύτερο. Ε, με χαρά λοιπόν θα ήθελα να καλωσορίσω τον Επίτροπο σε Julian King Θα ήθελα με την ευκαιρία αυτή να εκφράσω την συμπάθεια του συνόλου της Επιτροπής μας, των μελών της Επιτροπής μας σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδιαίτερα το Ηνωμένο Βασίλειο που υποφέρει από τις τελευταίες τρομοκρατικές ενέργειες. Γενικά εκδίδουμε συνήθως ανακοινώσεις σε σχέση με, αυτή τη, με αυτές τις ενέργειες, αλλά η σειρά των τρομοκρατικών ενεργειών σε όλο τον κόσμο, όχι μόνο στη δική σας χώρα, μας αναγκάζει σαν Ευρωπαϊκή Ένωση να είμαστε έτοιμοι να συνεργαζόμαστε με τις γειτονικές χώρες και με χώρες και δυνάμεις που έχουν μακροπρόθεσμη γνώση καταπολέμησης της τρομοκρατίας έτσι ώστε να γίνουμε όσο πιο ε, ανθεκτικοί ε, μπορούμε. Ξέρω ότι δεν έχετε πάρα πολύ χρόνο στην διάθεσή σας και γι' αυτό θα ήθελα κύριε Επίτροπε να σας δώσω το λόγο. Σας ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας. Χαίρομαι που έχω την ευκαιρία να ξεκινήσω με έναν διάλογο ο οποίος ελπίζω ότι θα συνεχιστεί με τα μέλη της Επιτροπής σας. Συμφωνώ πλήρως με τις τελευταίες παρατηρήσεις τις οποίες κάνατε, ότι δηλαδή στον τομέα αυτό, στα θέματα αυτά, δεν θα πρέπει να λειτουργήσουμε με, με περιορισμένο τρόπο θα έλεγα, οι ε, προκλήσεις τις οποίες αντιμετωπίζουμε και σε επίπεδο τρομοκρατίας και σε επίπεδο κυβερνοτρομοκρατίας προέρχονται από περιοχές εκτός της Ένωσης και εκδηλώνονται ε, σε ένα, εξελίσσονται σε μία μορφή απειλή την οποία θα χαρακτήριζα σαν πολυεθνική. Uh, uh, Γι' αυτό νομίζω ότι έχουμε να... Ευτυχώς είχαμε χτες εδώ στο Βέλγιο ε, μια αποτυχημένη απόπειρα. Αυτή η βομβιστική ενέργεια στην Γκάρ Σοντράλ ήταν η πέμπτη ε, τρομοκρατική ενέργεια μέσα σε λιγότερο από μήνα. Μάντσεστερ, Λόντον Bridge. Finsbury Park και Παρίσι. Συνεπώς λοιπόν έχουμε να κάνουμε με ένα ιδιαίτερα αυξημένο ρυθμό ε, ε, από τέτοιου είδους τρομοκρατικές ενέργειες, ο οποίος φαίνεται να αυξάνεται συνεχώς. Υπάρχει φυσικά αύξηση του επίπεδου ασφαλείας στις διάφορες χώρες ε, και θα συνεχιστεί η κατάσταση αυτή. Το ΤΑΕΣ πιέζεται επί τόπου στην Ανατολική Συρία και γι' αυτό αυξάνει τις εκκλήσεις για τέτοιου είδους τρομοκρατικές ενέργειες σαν αντίπεινα κατά κάποιο τρόπο και ζητούν να υπάρξουν επιθέσεις απέναντι, εναντίον των λεγόμενων soft στόχων νέων αθώων γενικά οι οποίοι ε, ε, συγκεντρώνονται σε συγκεκριμένες περιοχές. Αυτές οι ενέργειες ε, είναι εμπνευσμένε από τον τζιχαδισμό. Βλέπουμε δυστυχώς και κάποιες αντιδράσεις σε τέτοιου είδους. Αυτό που συνέβη στο Finsbury Park που γνωρίζω καλά στο Λονδίνο ήταν μια ισλαμοφοβική ενέργεια εις βάρος των μουσουλμάνων με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο το ΝΤΑΕΣ ζητά από τους πιστούς να χτυπήσουν τις υπόλοιπες κοινότητες. Η, θα έλεγα η διάκριση που γίνεται μερικές φορές ανάμεσα στις εσωτερικές και εξωτερικές πολιτικές ε, δυστυχώς όσο περνάει ο καιρός γίνεται ιδιαίτερα θεωρητική αυτό το οποίο είναι εξωτερικό τη μία, την επομένη δυστυχώς έχει καταστεί κάτι το διεθνές και εξωτερικό. Εμείς ήδη στα πλαίσια της συνολικής στρατηγικής του 2016 και της ατζέντα για την ασφάλεια το 2015 απαιτεί να υπάρξει μια ολοκληρωμένη από κοινού αντίδραση χρησιμοποιώντας όλα τα διαθέσιμα μέσα χρησιμοποιώντας την αμοιβαία βοήθεια, συνεργασία με βάση τις αξίες μας. Η ασφάλεια και η λειτουργική ασφάλεια είναι στόχος της Επιτροπής μας εξ αρχής. Ε, δημιουργήθηκε άλλωστε από τον κύριο Γιούνκερ ε, και ε, η θέση του Επιτρόπου για θέματα ασφάλειας, την οποία καλύπτει ο υποφαινόμενος, ε, και υπάρχουν υπηρεσίες, 20 γενικές διευθύνσεις ε, και άλλες υποϋπηρεσίες και τμήματα μεταξύ των οποίων και η υπηρεσία εξωτερικής δράσης που συνεργάζονται έτσι ώστε να υποστηρίξουν τις χώρες μέλη στον τομέα της ασφάλειας. Η εφαρμογή αυτής, ε, αυτού του προγράμματος για την ασφάλεια θα απαιτήσει μια αποτελεσματική και συνολική αντιμετώπιση όχι μόνο στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά σε όλα τα όργανα και σε αυτό εδώ το σώμα και θα συνεχίσουμε την προσπάθεια σε συνεργασία μαζί σας και τα άλλα όργανα μεταξύ των οποίων και με άλλους οργανισμούς όπως το ΝΑΤΟ. Να αναφέρω τώρα κάποιους από τους τομείς τους οποίους θα πρέπει να λειτουργήσουμε με συλλογικό τρόπο σε επίπεδο εσωτερικό και εξωτερικό. Καταρχάς σε θέματα τρομοκρατίας. Όπως ξέρετε την Δευτέρα το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων υιοθέτησε τις συστάσεις για την καταπολέμηση της εξωτερικής τρομοκρατίας έτσι ώστε οι αντιτρομοκρατικές μας δράσεις και ενέργειες να συνεισφέρουν στη μείωση της απειλής την οποία υφιστάμεθα στην παρούσα στιγμή. Τους προηγούμενους 18 μήνες πετύχαμε κάποια, κάποιους από τους στόχους αυτούς μέσω των διαλόγων για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας με τρίτες χώρες και της στήριξης που δώσαμε στις χώρες αυτές. Εμείς αποφύγαμε και αποτρέψαμε ενέργειες λοιπόν, εμείς στείλαμε εμπειρογνώμονες σε πάρα πολλές χώρες και οι ενέργειες αυτές θα ενισχυθούν σε συγκεκριμένους κατά προτεραιότητα τομείς όπως τα Δυτικά Βαλκάνια, η Τουρκία και η Βόρεια Αφρική. Υπάρχουν οι εξωτερικές υπηρεσίες όπως ε, η Europol, η Ευρωπαϊκή Ακτοφύλακη, ε, η ΣΥΠΑΛ, η ε, Eurojust επίσης βοηθούν τις χώρες στο τομέα της καταπολέμησης της τρομοκρατίας και θα πρέπει να βρούμε τρόπους βελτίωσης της συνεργασίας αυτής, λαμβάνοντας υπόψη βέβαια ότι οι χώρες δεν έχουν και άπειρους πόρους η συνεργασία ανάμεσα στις αποστολές ΚΕΠΑ, τύπου ΚΕΠΑ και τις υπηρεσίες που ασχολούνται με θέματα δικαιοσύνης και αστυνόμευσης θα ενισχυθούν στο μέλος. Η συλλογή στοιχείων από τις αποστολές της ΚΕΠΑ στα πλαίσια της τακτικής τους δραστηριότητας θα μπορούσε να περιλαμβάνει πληροφορίες για μεμονωμένους τρομοκράτες, για τα μόντους οπεράντι τους, ε, για τις μετακινήσεις τους ε, και για τους πόρους που έχουν στην διάθεσή τους. Τα στοιχεία αυτά θα είναι πολύτιμα για τις δικές μας κοινοτικές και εθνικές αρχές και θέλουμε να υπάρχει κυκλοφορία ε, της ενημέρωσης αυτού του τύπου. Εμείς προσπαθούμε λοιπόν να προωθήσουμε την συνεργασία και στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πέραν των σύνορων μας. Υπάρχει το δίκτυο συνειδητοποίησης της ριζοσπαστικοποίησης, είναι κάτι το οποίο υποστηρίζεται και από εμπειρογνώμονες στην Τουρκία, στα Δυτικά Βαλκάνια και την Τινησία. Εμείς θα διπλασιάσουμε την χρηματοδότηση για την καταπολέμηση των βίαιων τρομοκρατικών συμπεριφορών σε όλες αυτές τις περιοχές σε σχέση με το 2015. Έχουμε όμως ανάγκη από περαιτέρω πρόοδο μαζί με τους εταίρους μας έτσι ώστε να καταπολεμήσουμε τον εξτρεμισμό και την ριζοσπαστικοποίηση ιδιαίτερα στις, στα σοφρονιστικά ιδρύματα, στην καταπολέμηση της προπαγάνδας που χρησιμοποιείται ε, στο διαδίκτυο. Ε, ε, ασχολούμεθα λοιπόν με το φόρουμ της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το διαδίκτυο και μετά από την συνάντηση της ομάδας των 7 και την συνάντηση τον επόμενο μήνα της κορυφής της ομάδας των 20 θα πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι οι παροχής υπηρεσιών στο διαδίκτυο θα αυξήσουν τους ελέγχους τους για να μπλοκάρουν τις ακραίες συμπεριφορές και καταχωρήσεις και να προωθήσουν το σύστημα της αυτοματοποιημένης διαγραφής σελίδων. Να μπορούν δηλαδή με τρόπο μηχανικό να εντοπίζουν και να διαγράφουν συγκεκριμένα στοιχεία ενημερώνοντας το κοινό ότι προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε αυτήν την απαράδεκτη προπαγάνδα. Αυτό σε καμία περίπτωση δεν θέτει σε αμφισβήτηση το δικαίωμα στην ελεύθερη έκφραση, αυτή είναι βασική μας αξία στην οποία πιστεύουμε, αλλά είναι θέμα προστασίας των ευάλωτων τμήματων της κοινωνίας η οποία επέφτει θύμα αυτής της ύπουλης προπαγάνδας. Και αυτό θα πρέπει να συνοδεύεται βέβαια και από προσπάθειες στις ίδιες τις χώρες όπως και στα νοτιοδυτικά Βαλκάνια και στις αραβικές χώρες. Θα πρέπει να δημιουργήσουμε ένα νέο αφήγημα αν θέλετε το οποίο να δείχνει στις κοινωνίες τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα αυτό. Οι τρομοκράτες χρειάζονται χρήματα για την χρηματοδότηση των ενεργειών τους και η θα έλεγα διαταραχή αυτών των δικτύων, αυτών των διάβλων χρηματοδότησης θα επιτρέψει να μειωθεί ε, ο πλούτος αυτός και αυτό θα ωφελήσει θα έλεγα την δράση μας και τους στόχους μας. Φυσικά συνεργασία τεχνική με τις τρίτες χώρες, ανταλλαγή ενημέρωσης και πληροφοριών, εφαρμογή του Συμβουλίου των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας, όπως επίσης και εφαρμογή των διατάξεων για την καταπολέμηση του βρώμικου χρήματος. Σαν παράδειγμα, 16 εκατομμύρια για το ΜΕΝΑ και τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας έτσι ώστε να καταπολεμηθούν εκεί τα δίκτυα ξεπλήματος χρήματων. Ε, όλα αυτά είναι κρίσιμα για να ανοιχνεύσουμε, προλάβουμε και να παρεμποδίσουμε τη δράση των ομάδων αυτών είναι τμήμα θα έλεγα στήριξη των χωρών να ενισχύσουν και την ποινική τους δικαιοσύνη και τέλος <clears throat> το λαθρεμπόριο όπλων, ιδιαίτερα στα Δυτικά Βαλκάνια, είναι μια βασική προτεραιότητα. Θα πρέπει να γίνουν περισσότερα, να χρησιμοποιήσουμε τις εμπειρίες που έχουμε από τις συναντήσεις στον τομέα της δικαιοσύνης και της αστυνόμευσης ε, ε, μέχρι τώρα, για να καταπολεμήσουμε ακόμα περισσότερο το λαθρεμπόριο αυτό. Η άλλη απειλή αν θέλετε, την οποία έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι οι κυβερνοεπιθέσεις. έρχεται από κρατικές και μη κρατικές υπηρεσίες. Δυστυχώς διαπιστώνουμε ότι υπάρχει επιθυμία και ικανότητα δυστυχώς να χρησιμοποιείται ο κυβερνοχώρος για εγκληματικές δραστηριότητες και για λόγους πρόκλησης προβλημάτων σε άλλους και ε, για λόγους προπαγάνδας. Οι απειλές αυτές, ε, οι κεβέρνοαπειλές αν θέλετε, αυξάνονται και σε συχνότητα και σε κλίμακα. Θυμηθείτε ε, πριν λίγες εβδομάδες μια επίθεση στους υπολογιστές 150 χωρών σε όλο τον κόσμο. Αποτελεσματική δράση εναντίον όλων αυτών των απειλών απαιτεί μια σωστή προετοιμασία και συνεργασία. Γι' αυτό θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε τις τρίτες χώρες οι οποίες θα πρέπει να βελτιώσουν τις ε, δυνατότητες αντίδρασης και ανθεκτικότητας σε κυβερνοεπιθέσεις όπως επίσης και διερεύνηση των υποθέσεων αυτών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην παρούσα φάση αναθεωρεί ε, την στρατηγική η οποία ε, αποφασίστηκε το 2013 και τα πράγματα αλλάζουν πια πολύ γρήγορα και βασικός μας στόχος είναι και να μειώσουμε τις ε, δυνατότητες επιθέσεων τέτοιου είδους αλλά και τις συνέπειές τους όταν υπάρχουν τέτοιου είδους επιθέσεις. Δεν είναι μόνο πρόληψη δηλαδή αλλά ανείχνευση και αποτροπή ε, και επίσης θέλουμε να υπάρχει διεθνής εμπλοκή με άλλους κομβικούς εταίρους και διεθνείς οργανώσεις. Το δίκτυο των διεθνών σχέσεων το οποίο έχουμε αναπτύξει είναι κεντρικό για την υπόθεση αυτή. Είναι προϋπόθεση ε, για την επιτυχία της προσπάθειας που κάνουμε σε συνεργασία με τους στρατηγικούς εταίρους μας στις Ηνωμένε Πολιτείες ιδιαίτερα. Εγώ με τον Δημήτρη Αβραμόπουλο είχαμε πάει στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας στην συνάντηση για θέματα δικαιοσύνης ε, με τις Ηνωμένε Πολιτείε και ενημερωθήκαμε για τις προσπάθειες που κάνουν οι Αμερικανοί στα πλαίσια της καταπολέμησης της κυβερνοτρομοκρατίας. Συνεργαζόμαστε και με τον ΟΑΣΕ, την Ίντερπολ, τα Ηνωμένα Έθνη, την Διεθνή Ομάδα για την Καταπολέμηση της Χρηματοδότησης κτλ βασιζόμαστε στο πρόγραμμα δράσης το οποίο βασίζεται με τη σειρά του στην δήλωση την κοινή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ του Δεκεμβρίου του 2016 ε, στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων κατέληξε ε, σε αποφάσεις για την συνεργασία με το ΝΑΤΟ και για το πρόγραμμα δράσης έχει σημειωθεί πρόοδος και στον τομέα της κυβερνοασφάλειας και της άμυνας. Ε, το έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έγγραφο θέσεων προς επεξεργασία, ε, δείχνει ότι ανεξάρτητα από τον δρόμο που θα ακολουθήσουμε η στενή συνεργασία με το ε, Βορειοατλαντικό Σύμφωνο είναι καθοριστικός παράγων. Συνεπώς λοιπόν έτσι θα αντιμετωπίσουμε τις σοβαρές απειλές, αυτές τις διεθνικές απειλές της κυβερνοτρομοκρατίας και της τρομοκρατίας απαιτείται να υπάρξει συντονισμένη απάντηση, δεν πρόκειται από μόνες τους να αυτοαναιρεθούν οι απειλές αυτές και θα πρέπει σε έναν συνεχώς θα έλεγα αλληλοεπηρεαζόμενο κόσμο να συνδυάσουμε τις εξωτερικές και εσωτερικές μας πολιτικές. Θα πρέπει να διαμορφώσουμε μια ενιαία αντιμετώπιση του προβλήματος που να συνδυάζει τον εσωτερικό και εξωτερικό μας χώρο. Ε, σαν διπλωμάτης πιστεύω ότι είναι απαραίτητο να συνδυάσουμε την εμπειρία που έχουμε και την συνεργασία ανάμεσα στο εξωτερικό και το εσωτερικό κομμάτι και τότε θα έχουμε περισσότερες πιθανότητες να πετύχουμε. Νομίζω λοιπόν ότι με την δική σας συνδρομή θα μπορέσουμε να σημειώσουμε πρόοδο στο σύνολο των θεμάτων αυτών και προσβλέπω σε περαιτέρω συζητήσεις μαζί σας. Ευχαριστώ πολύ για την ε, παρέμβασή σας και θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στους συναδέλφους μου για να θέσουν ερωτήσεις ή να υποβάλουν παρατηρήσεις. Κύριε Φρόιντ, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και ευχαριστώ και σας Τζούλιαν για την προσέλευσή σας και θα ήθελα να σας ε, πιστήσω την προσοχή σε ένα θέμα που είναι ουσιώδες αλλά δεν έχει θυγεί ακόμη. Τουλάχιστον είναι ουσιώδες από ό,τι το βλέπω εγώ. Και εννοώ την ενδεχόμενη κυβερνοεπίθεση στο Power Group της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι μια επιχείρηση υβριδικού χαρακτήρα στην Ουκρανία από τη Ρωσία από ό,τι φαίνεται. Ψάξαν να δούνε δηλαδή ένα είδος, σε ένα είδος πειραματισμού τι μπορούν να κάνουν σε ολόκληρη σχεδόν τη χώρα για να ρίξουν εντό εισαγωγικών την παροχή ενέργειας. Διερωτώ με πώς, τι επιπτώσεις μπορεί να έχει αυτό σε ευρύτερο πλαίσιο, όπως είναι ολόκληρη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Διερωτώ με αν μπορείτε να απαντήσετε σε κάποιες ερωτήσεις σχετικά. Πόσο ανησυχείτε, ότι αυτό μπορεί να είναι η επόμενη φάση του τι μπορεί να συμβεί εδώ στην Ευρώπη. Τι είδους αντίμετρα συζητούνται για την πρόληψη τέτοιου ενδεχομένου. Και υφίσταται συνεργασία με τον ε, συνεπίτροπό σας κύριο Σεύκοβιτς που έχει το χαρτοφυλάκι για την ενέργεια και έχετε και κάποια συμβουλή για το τι μπορεί να συμβεί σε περίπτωση μακροχρονιότερης διακοπής ρεύματος και βέβαια δεν θα είναι απαραίτητα να γίνει σε μία μέρα όπως η σημερινή που θα καθίσουμε εδώ χωρίς ρεύμα και μπορεί να μην κρατήσει μόνο μία μέρα αλλά, αλλά ίσως και μία εβδομάδα και περισσότερο. Εσείς κύριε Τάνοκ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε. Θα ερωτήσω σχετικά με τη δική μας χώρα, αν και αντιλαμβάνομαι ότι είναι δύσκολη θέση σας. Έχω δύο ερωτήσεις. Μία αφορά την έναρξη χθες των διαπραγματεύσεων για το Brexit, όπου σαφώς το Ηνωμένο Βασίλειο αποδέχεται διστακτικά δύο φάσεις και τα θέματα ασφαλείας φαίνεται πως θα συζητηθούν και όλα τα ε, σχετικά με JAI, με εσωτερικά και ασφάλεια, στοιχεία επιβατών, SIS και ούτω καθεξής, θα ε, αρχίσουν να συζητούνται μάλλον του χρόνου. Σας ικανοποιεί αυτό. Και είστε πεπισμένος ότι δεν υπάρχει, θα έχετε διαβάσει το έγγραφό μου, ότι βρισκόμαστε στο χείλος του γκρεμού. Και βεβαίως από την άλλη μεριά όλοι λένε ότι τίποτε δεν έχει συμφωνηθεί, αν δεν συμφωνηθούν όλα και προχωρώντας για να συμφωνήσουν πέφτουν τελικώς στον κρεμό. Και έχω και μια άλλη ερώτηση πάλι σχετικά με το Ηνωμένο Βασίλειο. Μιλήσατε για την τρομοκρατική επίθεση στο Μάντσεστερ. Η Πρωθυπουργό κυρία Μέη σχολίασε την επόμενη μέρα ότι θα χρειαστεί να διεξαγάγουμε δύσκολε συζητήσει με ορισμένου από του φίλου μα. Εγώ το ερμηνεύω αυτό ω ότι εννοεί χώρες όπως η Σαουδική Αραβία και το Κατάρ και ότι θα πρέπει να τους πούμε στο μέλλον ότι είναι απολύτως απαράδεκτη η κατάσταση του να χρηματοδοτούν τσιχατιστικά κινήματα στη Συρία και αλλού, τα οποία έχουν τώρα και ένα spill-over effect και ριζοσπαστικοποίηση και επιθέσει τελικώς στη δική μας χώρα. Και βεβαίως και την αντιπαράθεση πρόσφατα μεταξύ Σαουδαράβων και Κατάρ, το οποίο Κατάρ έχει τεράστιες επενδύσεις και στη Σαουδική Αραβία αλλά και στο Λονδίνο και επενδύουν ό,τι μπορούν στο Λονδίνο, στο Ηνωμένο Βασίλειο και μερικά από τα λεφτά αυτά είναι, πληρώνονται και ως λίτρα στην Αλκάιδα για την απελευθέρωση στελεχών τους. Κάνουμε τέτοιες δύσκολες συζητήσεις με τους φίλους μας. Είπε η Πρωθυπουργός κυρία Μέη ότι θα καταστήσω απολύτως σαφές ότι είναι απαράδεκτο για μας να ε, χρησιμοποιούν τα χρήματά μας με τέτοιο τρόπο. Δηλαδή η απόδοση των κεφαλαίων που επενδύουν στο Ενωμένο Βασίλειο. Φώτιγκα, δύο ερωτήσεις. Παρακολουθήσαμε πριν την παρουσίαση μελέτης από δύο εμπειρογνώμονες του ISS, την κυρία Γκάουπ και την κυρία Πάουελς, Μερικές από τις παρατηρήσεις που έκαναν ε, ήταν πραγματικά πάρα πολύ ανησυχητικές από αυτές που ακούσαμε δηλαδή σχετικά με το επίπεδο συνεργασίας μεταξύ χωρών στη νότια γειτονιά μας σε ό,τι αφορά τον εντοπισμό τρομοκρατών, τις δραστηριότητε τους κλπ. Αυτά που είπατε και εσείς και τα ονομάσατε travel patterns είναι πιθανότερο να υπάρξει συνεργασία με ευρωπαϊκούς θεσμούς, είτε ξεχωριστά σε διπερές δηλαδή επίπεδο, παρά να καταλήξουν από κοινού σε κάποια συμφωνία. Και γνωρίζουμε ότι η τρομοκρατία δεν γνωρίζει σύνορα. Δεύτερο, σε ό,τι αφορά το ξέπλυμα του βρώμικου χρήματος, όταν πήγε η υποεπιτροπή μας αποστολή για να παρακολουθήσει την αποστολή της Σοφία στη Ρώμη, John F. Formed, μιλήσαν εκεί για επενδύσεις, investing patterns, λαθοδιακινητών μεταναστών που χρησιμοποιούνται για διαφόρους σκοπούς. Το ίδιο συνέβη και με τους πειρατές στο κέρας της Αφρικής και αλλού. Ορισμένες από αυτές τις διαδρομές των ε, τρομοκρατών είναι παρόμοιες με αυτού, ακολουθούν δηλαδή τους ίδιους οδούς με το οργανωμένο έγκλημα. Με ποιους τρόπους μπορεί να, να οργανωθεί μια συνεργασία με τις χώρες της νότιας γειτονίας, αλλά και περαιτέρω και προς Ανατολάς και προς Νότον έτσι ώστε να ξεριζωθεί αυτό το κακό. Ο κύριος Νάρτ. Precisamente Θα ήθελα να αναφερθώ σε κάτι που είπατε εσείς, κύριε Πρόεδρε. Το οργανωμένο έγκλημα δεν μπορεί να λειτουργήσει και να είναι αποτελεσματικό χωρίς ε, στήριξη και διοικητική μέρημνα. Γνωρίζω πολύ καλά αυτό το θέμα γιατί ήμουν δικηγόρος, ε, ποινικό ήταν ε, κυρίως ποινικό ήταν ο που με απασχόλησε και ασχολήθηκα ιδιαίτερα και με τους φορολογικούς παραδείσους. Ξέρουμε ότι οποιοδήποτε θέλει να είναι αποτελεσματικός κατά του οργανωμένου εγκλήματος θα πρέπει να διαλευκάνει όλες τις διαδικασίες και τα κανάλια που χρηματοδοτούν την εγκληματική αυτή δραστηριότητα και που βοηθούν να διοχετευθούν καθόπιν τα κονδύλια στους φορολογικούς ε, παραδείσους. Οι επαφές λοιπόν και οι διασυνδέσεις μεταξύ της ε, διακίνησης παράνομων ουσιών, ναρκωτικών, και του οργανωμένου εγκλήματος, οι διαδρομές που ακολουθούν τα χρήματα, όλοι αυτοί παραδείγματος χάρη που έχουν λογαριασμούς σε τράπεζες που βρίσκονται σε αυτές τις περιοχές. Η φοροαποφυγή, η χρήση φορολογικών παραδείσων όπως οι Βερμούδες, τα νησιά Καϊμάν, είναι καθοριστικό να διαλευκανθούν. Δεν υπάρχει περίπτωση, αν δεν έχουμε τις πληροφορίες για όλα αυτά, να μπορέσουμε να είμαστε αποτελεσματικά. Και χειρίζονται δράσεις παρόμοιες με αυτό που έγινε με το Panama Paper. Πέρα λοιπόν από τους φορολογικούς ε, παραδείσους, πέρα από την στήριξη και τη χρηματοδότηση αυτής της ε, εγκληματικότητας, θα πρέπει να υπάρξει και μία χρηματοδότηση συνεργασίας μεταξύ των χωρών. Ναι, η Ολλανδία παραδείγματος χάρη. Τι ρόλο παίζει όσον αφορά τις φορολογικές έδρες, τις δηλώσεις. Ξέρουμε πολύ καλά ότι δεν είναι απλό να βρει κανείς την αλήθεια. Well, no Δεν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις. Κύριε Πίτροπε μπορείτε να απαντήσετε ή να εκφράσετε τις σκέψεις όσον αφορά αυτό που ακούσαμε. Ε, ε, Disculpe, Σας ζητώ συγγνώμη. Θέλω να ξαναπάρω το λόγο. Για να πω ότι η τρομοκρατία οι τζιχαντιστές. Δεν μπορούμε να τους καταπολεμήσουμε αν δεν υπάρξει ανταλλαγή πληροφοριών. Ειλικρινά λοιπόν, εάν στην Ευρώπη δεν υπάρχει εμπιστοσύνη μεταξύ των ε, υπεύθυνων στις υπηρεσίες πληροφοριών, εάν δεν θεωρούμε ότι οι εταίροι μας δεν είναι αξιόπιστοι, γιατί αυτό ακούμε ε, off βέβαια όταν ε, ζητήσουμε την άποψη κάποιων ειδικών στον τομέα των πληροφοριών. Εάν λοιπόν δεν υπάρχει αξιοπιστία κάποιων χωρών στη Νότια Μεσόγειο, πώς μπορούμε να συνεργαστούμε αποτελεσματικά μαζί τους. Ναι, τώρα καταλαβαίνω, λέει η Πρόεδρος. Μπορώ λοιπόν να δώσω το λόγο στον Επίτροπο. Uh, ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ γιατί βλέπω ότι σας αφορά πολύ το θέμα αυτό. Θα προσπαθήσω να παρουσιάσω τα θέματα τα οποία θίξατε. Αν δεν απαντήσω σε κάτι από αυτά που θίξατε, μπορείτε να επανέλθετε. Καταρχήν, ποια είναι η δράση μας ε, για την καταπολέμηση του κυβερνοεγκλήματος, τι κάνουμε στον κυβερνοχώρο και ιδιαίτερα για την προστασία υποδομών ζωτικής ε, σημασίας, όπως δίκτυα μεταφορών ε, ή άλλα σημαντικές ε, υποδομές. Προσπαθούμε να μάθουμε από τις πρόσφατες επιθέσεις και έχετε δίκιο όταν λέτε ότι το πολύ ενδιαφέρον άρθρο που δημοσιεύτηκε αυτήν την εβδομάδα εξάλλου για τις επιθέσεις στην Ουκρανία κατά το τομέα της ενέργειας, των υποδομών ε, στον τομέα της ενέργειας. Χρησιμοποιείται λοιπόν εδώ ο κυβερνοχώρος και υπάρχουν συγκεκριμένες επιπτώσεις στον πραγματικό μας κόσμο. Και στην Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν και στο ΝΑΤΟ έχουν ε, επεξεργαστεί το θέμα αυτό και το σκεφτόμαστε πολύ σοβαρά από την άποψη τη δική μας, η Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουμε αποφασίσει να ξεκινήσουμε έναν πολύ ειλικρινή διάλογο μεταξύ ημών των κρατών μελών και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά το θέμα αυτό, όσον αφορά την αύξηση παραδείγματος χάρη της αποτροπής προς όλους αυτούς που θέλουν να χρησιμοποιήσουν τον κυβερνοχώρο για να επιτεθούν. Και μεταξύ της ε, επεξεργασίας αυτής, η οποία θα διαρκέσει μέχρι το Σεπτέμβριο, και των προτάσεων που θα υποβάλουμε τον ε, το φθινόπωρο, πιστεύω ότι θα είμαστε σε θέση να υποβάλουμε μια βάση προσυζήτηση που θα συμπεριλαμβάνει ουσιαστικά τις δυνατότητες ε, τις οποίες θέλουμε να ενισχύσουμε όσον αφορά την προστασία των υποδομών μας, όσον αφορά τη δυνατότητα ανταπόκρισης, αντίστασης. Σαφώς και θα πρέπει να ενισχύσουμε το ΕΝΙΣΑ, τη δυνατότητα δημιουργίας ομάδων για την αντιμετώπιση κρίσεων, και θα πρέπει βεβαίως να αναλύσουμε κάποια παραδείγματα που διαθέτουμε διεθνώς. Στις Ηνωμένες Πολιτείες παραδείγματος χάνει υπάρχει ένας πολύ συγκεκριμένο μοντέλο συνεργασίας για την προστασία και την αντιμετώπιση υποδομών ζωτικής συμμαχίας μεταξύ του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα. Έχουμε αυτό το παράδειγμα αλλά και κάποια άλλα. Θα πρέπει λοιπόν να ξεκινήσει μια μεγάλη συζήτηση για όλα αυτά τα θέματα καθώς και για τη βελτίωση της συνεργασίας μας, της συνεργασίας ανάμεσα στον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα. Και βεβαίως ε, ο ιδιωτικός τομέας που παίζει ένα καθοριστικό ρόλο σε όλες αυτές τις ε, υποδομές ζωτικής σημασίας και θα πρέπει να στηρίξουμε οι δε, να μοιραστούμε πληροφορίες και να επενδύσουμε από κοινού σε έρευνα για να βελτιωθεί η ασφάλεια. Η πρώτη εταιρική σχέση δημόσιου και ιδιωτικού τομέα με επιδότηση 2 δισεκατομμύριων ευρώ από φασίστηκε για την περίοδο 2017-2021 προστασία υποδομών ζωτικής συμμαχίας και όπως ε, σας είπα, αυτό είναι κάτι που γίνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μόνο για το 2017 οι επενδύσεις φτάνουν το ποσό των 19 δις. Καταλαβαίνετε ότι απέχουμε πολύ από τις Ηνωμένε Πολιτείες. Πρέπει λοιπόν να κινητοποιηθούμε, να αυξήσουμε τις προσπαθειές μας, γιατί οι προκλήσεις είναι πολύ σημαντικές. Παράλληλα με αυτήν την στρατηγική εξετάζουμε και άλλους τομείς που άπτονται του τομέα της ενέργειας, που είναι καθοριστικοί. Και βεβαίως εδώ θα πρέπει να δούμε και κάποιες συμπεριφορές. Συχνά και εμείς οι ίδιοι έχουμε συμπεριφορές που αφήνουν κενά, που επιτρέπουν κάποιες αδυναμίες και δημιουργούν αδύναμα σημεία. Γι' αυτό και μεταξύ ημών των ε, εταιριών που ενεργοποιούνται στον τομέα της πληροφορικής, των φορέων παροχής υπηρεσιών στο διαδίκτυο, θα πρέπει να συνεργαστούμε για να βελτιώσουμε την ασφάλεια των δικτύων και των συστημάτων πληροφορικής. Χρειάζεται επίσης και διεθνή συνεργασία και αυτό σημαίνει όχι απλώς να συνεργαστούμε με χώρες που σκέφτονται όπως και εμείς, αλλά τουλάχιστον να ξεκινήσουμε συζήτηση με χώρες οι οποίες σκέφτονται διαφορετικά από εμάς για τα θέματα αυτά. Την Κίνα και τη Ρωσία παραδείγματος χάρη. Μπορεί να μην μπορέσουμε να συνεργαστούμε ευρύτατα ακόμα με τις χώρες αυτές, αλλά σίγουρα υπάρχουν κάποιοι στην Κίνα και στη Ρωσία που έχουν εκφράσει την απεσιοδοξία τους, τη δυσαρέσκειά τους καθότι αυτές οι δραστηριότητες πολλές φορές προέρχονται από τις χώρες αυτές. Θα μπορέσουμε ίσως λοιπόν να ξεκινήσουμε μια συζήτηση με αυτούς οι οποίοι έχουν εκφράσει αυτές τις ανησυχίες και τη δυσαρέσκεια για να περιορίσουμε τις επιθέσεις των κυβερνοχώρα που προέρχονται από τη Ρωσία και την Κίνα. Ξεκινάμε λοιπόν μια συζήτηση με τις χώρες μέλη και πιστεύω ότι θα είμαστε έτοιμοι να υποβάλουμε προτάσεις μέχρι το φθινόπωρο. Για το Brexit τώρα και την εξωτερική πολιτική της Μεγάλης Βρετανίας. Εγώ δεν εκπροσωπώ πλέον, όπως ξέρετε, την κυβέρνηση της αυτού μεγαλειότητας. Όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις τώρα για το Brexit, Νομίζω ότι ο Μισελ Μπαγνιέ, η ομάδα του, οι συνεργάτες του θα είναι αυτοί που θα μπορέσουν να σα απαντήσουν ε, στις ερωτήσει που έχετε. Όταν φτάσουμε στο στάδιο αυτό των διαπραγματεύσεων και φτάσουμε στη συζήτηση για το μέλλον της κοινή μας ασφάλειας και τα θέματα που από το ασφάλειες, βεβαίως και εγώ θα μπορέσω να εκφράσω τις απόψεις μου και τις προτάσεις μου και πιστεύω ότι σαφώς και θα καλύψουμε καλύτερα τα θέματα της ασφάλειας με συνεργασία. Εάν λοιπόν η κυβέρνηση της Μεγάλης Βρετανίας υποβάλλει τις θέσεις της όπως το πρότεινε η Πρωθυπουργό η Τερέζα Μέη, εάν συνεχίσει η θέση αυτή να είναι στενή συνεργασία για θέματα ασφάλειας, εγώ βεβαίως θα στηρίξω τη θέση που ελπίζω να είναι η θέση της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης να βρούμε μια διαρθρωμένη συνεργασία ενίσχυσης της ασφάλειας για το μέλλον. Και πιστεύω ότι βεβαίως καταρχήν θα πρέπει να έχουμε κάποιους κοινούς στόχους, αλλά αυτό δεν αρκεί για να τους πετύχουμε. Θα είναι περίπλοκη η επεξεργασία των θεμάτων αυτών. Εξαρτάται και από τις θέσεις, επαναλαμβάνω, της Μεγάλης Βρετανίας. Και αυτό πιστεύω θα συμβεί πριν το τέλος του χρόνου ή στην αρχή του 2018. Έχουμε πάντως κοινό συμφέρον να μην υπάρξει χάσμα μεταξύ ημών και ημών και η έλλειψη συμφωνίας παραδείγματο χάρη όσον αφορά τα δεδομένα, την αντιστοίχηση βιομετρικών δεδομένων, τα συστήματα. Κανονικά το Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να αποκλειστεί από αυτές τις βάσεις δεδομένων. Αλλά πιστεύω ότι αυτό θα είναι σαφώς απώλεια και για την ασφάλεια του Ηνωμένου Βασιλείου, αλλά και για την ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να βρεθούν τρόποι να αποφευχθούν τέτοιες αποκλήσεις. Όσον αφορά τις χώρες του κόλπου, νομίζω ότι δεν είμαι αρμόδιος να απαντήσω. Θα πρέπει να απευθυνθείτε σε κάποιον που είναι αρμόδιος. Εμείς και στα πλαίσια της συνεργασίας μας με χώρες της Μέσης Ανατολής, στα διάφορα όργανα συνομιλιών και συνεργασίας, έχουμε αυξήσει τις προσπαθίες μας για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και της βίας. Αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις αυτές, προσπαθώντας να αντιμετωπίσουμε τη βία και την τρομοκρατία στις χώρες αυτές, να καταπολεμήσουμε όμως και τον εξτρεμισμό και τη βία και τη βία έκφρασή του και στις δικές μας χώρες. Και με το διάλογο και την συνεργασία με κάποιες από τα όργανα αυτά στα οποία συμμετέχουν οι χώρες του κόλπου πιστεύω ότι είναι το κατάλληλο φόρουμ για να ενισχύσουμε τη συνεργασία μας. Όσον αφορά τώρα την νότια πολιτική γειτονία μας, βεβαίως, εδώ οι σχέσεις με τις χώρες αυτές δεν είναι πάντα δεν είναι πάντα οι πιο εύκολοι συνομιλητές. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να θέσουμε στόχους, να επεξεργαστούμε τη συνεργασία μας και τα συμπεράσματα που πήραμε τη Δευτέρα στο Συμβούλιο είναι ένα βήμα για να προχωρήσουμε ακόμα παρετέρω στην διαρθρωμένη συνεργασία. Πολύ συχνά η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκίνησε αυτό το διάλογο για την καταπολέμηση της ε, τρομοκρατίας και μάλιστα προτείναμε να την καθώσουμε εμείς. Αλλά κατά κάποιο τρόπο ο σχεδιασμός που κάναμε δεν αντιστοιχούσε σε αυτό που μπορούσε και επιθυμούσε να κάνει η χώρα με την οποία συνεργαζόμαστε και θα πρέπει σαφώς να αλλάξουμε την πολιτική μας, να την προσαρμόσουμε στη χώρα με την οποία συνεργαζόμαστε. Η Λιβύη, παραδείγματο χάρη, είναι μια τελείως διαφορετική χώρα από άλλες με τις οποίες συνεργαζόμαστε. Πρέπει να έχουμε μια διαφορετική πολιτική με την ακτοφυλακή, να ενισχύσουμε τα νότια σύνορα της Λιβύης με την Τινησία και το Μαρόκο. Οι στόχοι είναι διαφορετική με την Αλγερία η οποία δεν είναι όσο ανεπτυγμένη θα ήθελε η ίδια να είναι η συνεργασία μας. Έχουμε βεβαίως λοιπόν κάποιες διαδικασίες, κάποιους κανόνες συνεργασίες με τις χώρες αυτές. Πρέπει όμως να λάβουμε υπόψη μας τους περιορισμούς των δικών τους συστημάτων, της δικαιοσύνης τους και το πώς οι ίδιοι μπορούν να προχωρήσουν σε αυτή τη συνεργασία. Τώρα, όσον αφορά την νομοποίηση πόρων από παράνομες δραστηριότητε, όσον αφορά τη διακίνηση, του διακίνητέ. νομίζω ότι έχει προβληθεί εξάλλου και μια συνάντηση κάπου εδώ σε αυτό το κτίριο για το θέμα αυτό των διακινητών. Αυτό είναι κάτι που σαφώς και πρέπει να γίνει αυτές οι δραματικές ε, ιστορίες οι οποίες συνεχίζονται θα πρέπει σαφώς να σταματήσουν. Είναι σαφές ότι κάποια από τα χρήματα αυτής της παράνομης δραστηριότητας χρηματοδοτούν τη τρομοκρατία. Και βεβαίως εμείς συνεχίζουμε τις προσπάθειές μας για να εντοπίσουμε τα κανάλια αυτής της χρηματοδότησης. Για το οργανωμένο έγκλημα, δεν μπορώ εγώ να μιλήσω εξ ονόματος ε, της κυβέρνησης της Μεγάλης Βρετανίας, ούτε της κυβέρνησης μπορώ να μιλήσω για το Γιβραλτάρ, αλλά σαφώς και στα διάφορα όργανα συνεχίζονται οι προσπάθειες για την εξάλληψη των δικτύων και το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, για να βρεθούν οι διασυνδέσεις με τους φορολογικούς παραδείσους και όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για μας. Και ένα ευρύ φάσμα μέτρων που γνωρίζετε έχουν ε, συμπεριληφθεί στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας ε, και του ξεπλήματος βρώμικου χρήματος Μία σειρά μέτρων λοιπόν που υλοποιούνται. Εναρμόνιση παραδείγματος χάρη των ε, ποινικών ε, κυρώσεων, οι παράνομες πληρωμές ε, με cash, καθώς και ό,τι αφορά την κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων και τις υπόλοιπες κυρώσεις που πρέπει να επιβάλλονται. Ανταλλαγή πληροφοριών. Θα ήθελα εδώ να κάνω κάποια σχόλια. Καταρχήν, υπάρχει ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών και αυτή συνεχίζεται και αυτό συμβαίνει και με άλλους σημαντικούς εταίρους μας όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες. Βεβαίως και χρειάζεται ενίσχυση αυτής της ανταλλαγής πληροφοριών και της συνεργασίας. Όσον αφορά τη βασική ε, βάση δεδομένων για την υποβολή του νόμου, είναι το σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών του Σέγγεν, το ΣΥΣ η δέσμευση των κρατών μελών για την ε, συμμετοχή στο δίκτυο αυτό αυξάνεται διαρκώς τα τελευταία χρόνια και το 2016 μόνο οι πληροφορίες για θέματα που αφορούν τρομοκρατία, εγκληματικέ δραστηριότητε, αυξήθηκε κατά 40%. Τα κράτη-μέλη, λοιπόν, βλέπουμε, συμμετέχουν, χρησιμοποιούν και μοιράζονται πληροφορίε βάσει αυτού του συστήματος και μέσω αυτού του συστήματος, καθότι έχουν διαπιστώσει ότι είναι χρήσιμο και νιώθουν, όπως είπαμε και στην αρχή, ότι η αύξηση αυτών των επιθέσεων με ταχύτατους ρυθμούς έχει οδηγήσει τα κράτη-μέλη σε μια μεγαλύτερη συμμετοχή και ανταλλαγή πληροφοριών. Και βεβαίως όσον αφορά τις πληροφορίες θα πρέπει να πούμε ότι δεν είναι σωστό ότι δεν λειτουργούν τα δίκτυα. Υπάρχει ε, ένα ευρωπαϊκό δίκτυο για την ανταλλαγή πληροφοριών. Αυτό λειτουργεί και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει ενισχυθεί πρόσφατα, λειτουργεί. Υπάρχουν μάλιστα, όπως ξέρετε, και στην Ολλανδία τα κεντρικά γραφεία τα μέλη των μυστικών υπηρεσιών, των υπηρεσιών πληροφοριών από όλα τα κράτη-μέλη της Ευρώπης συμμετέχουν, βρίσκονται εκεί, διερευνούν από κοινού υποθέσεις, μοιράζονται πληροφορίες και λειτουργεί το σύστημα. Βεβαίως και δεν μπορώ εδώ να αναφερθώ σε συγκεκριμένες υποθέσεις, αλλά πιστεύω ότι είναι πολύ σωστό να ενημερώσουμε ότι υπάρχει αυτό το δίκτυο, ότι συμμετέχουν όλες οι χώρες και ότι είναι αποτελεσματικό. Η κυρία Φώτιγκα. Κρίμα που έχουν ε, και χρονικά όρια. Έχετε όμως και εσείς. Δηλαδή, αν, αλλιώς θα ήθελα να κάνω δύο ερωτήσει. Λέει η ίδια η πρόεδρος, η κυρία Φώτιγκα. Πρώτα, οι τρόποι συνεργασίας μεταξύ Ευρωπαϊκής ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης και στον, στην κυβερνοασφάλεια επίσης και στη διάρκεια της ανταλλαγής απόψεων με τον ε, πρέσβη κ. Πέδρο Σεράνο της Υπηρεσίας Εξωτερικών Δράσεων χώρες που είναι χώρες εταίροι και για τον ΝΑΤΟ και για την Ευρωπαϊκή Ένωση δηλαδή εννοώ τη Μορδαβία, Βοσνία, Ζεγοβίνη και την Ισία. Χρειάζεται να επεξεργαστούμε ειδικού τρόπους συνεργασίας με τις χώρες αυτές, country specific ways, διότι για δύο τουλάχιστον χώρες συζητήσαμε την ενδεχόμενη σχέση τους με τις εξελίξεις στα Δυτικά Βαλκάνια θα συζητήσουμε καθώς επίσης και την μικροχρηματοδοτική ενίσχυση στην Μολδαβία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να βοηθήσουμε όχι μόνο τη Βοσνία Ζεγοβίνη, αλλά και όλες τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων στην δική τους προσπάθεια καταπολέμησης των κυβέρνοεπιθέσεων και να ενισχύσουμε την ανθεκτικότητά τους σε θέσεις. Υπάρχει κάποιος τρόπος να περιβληθεί αυτό τη μορφή ενός πιλωτικού προγράμματος ή ενδεχομένως μιας εμβληματικής πρωτοβουλίας ε, σε ό,τι αφορά τη συνεργασία μεταξύ θεσμικών οργάνων. Και δεύτερο, μας μιλήσατε για μια οριζόντια συνεργασία με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς για ζητήματα τρομοκρατίας μεταξύ γενικών διευθύνσεων των διαφόρων χαρτοφυλακίων και με την Υπηρεσία Εξωτερικών Δράσεων τι είδου συνεργασία περιμένετε από επιμέρους χώρες μέλη. Το δίκτυο αυτό ε, μπορεί να διευρυνθεί ώστε να περιλάβει και χώρες μέλη. Για να διευκρινίσουμε λίγο το τελευταίο σημείο. Εγώ μιλώ για μια οριζόντια ομάδα ειδικών καθηκόντων, cross-cutting task force, που περιλαμβάνει υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της ε, Υπηρεσίας Εξωτερικών Δράσεων και της Γραμματείας του Συμβουλίου. Προφανώς από εκεί προέρχονται ιδέες και προτάσεις από τη συνεργασία αυτή που εξορισμού την υλοποίησή τους θα αναλάβουν οι χώρες μέλη διότι απαιτείται νομοθεσία και συνεργαζόμαστε με τις χώρες μέλη για την εφαρμογή και μάλιστα πολύ στενά. Δεν σημαίνει ότι οι χώρες μέλη συμμετέχουν στην, ε, στον φορέα αυτόν. Για την πρώτη σας ερώτηση για, τα, για τις και ούτω καθεξής, ως πρώτο βήμα, τρεις ε, πιλωτικές χώρες, Μολδαβία, Τινησία, Βοσνία, Ζεγοβίνη, προχωρούμε σε διερεύνηση των δυνατοτήτων συμφωνίας καθώς και σε επέκταση του δικτύου και προς Ανατολάς και προς, και προς Νότον μάλλον για να μπορέσουμε να ε, συμφωνήσουμε ειδικώ για, για θέματα κυβερνοχώρου πρέπει να βαθύνουμε την ε, συνεργασία μεταξύ ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης και μεταξύ των δύο αυτών και των τρίτων χωρών εταίρων. Και για να σας πω και την προσωπική μου άποψη, είναι και ένα από τα θέματα που θα θέλαμε να αναπτύξουμε μέσα στα πλαίσια της στρατηγικής επανεξέτασης των θεμάτων ε, κυβερνοχώρου με μια ευρεία προσέγγιση για μια κυβερνοαποτροπή που σημαίνει, βεβαίως εδώ υπάρχει και μια στρατιωτική διάσταση η οποία συζητείται σε ορισμένα Υπουργεία Αμήνης και μπορεί να συζητηθεί μάλιστα και περαιτέρω και στο ΝΑΤΟ αλλά είναι ένα ευρύτερο στοιχείο αποτροπής το οποίο συζητείται για εκτός Υπουργείων Αμήνης στα πλαίσια της επιβολής του νόμου και που μπορεί και θα πρέπει να συζητηθεί και, με, και μεταξύ των χωρών μελών για να μην επιτρέψουν στους εγκληματίες να ξεφύγουν διότι πρέπει να κληθούν υπόλογοι ενώπιον της δικαιοσύνης άνθρωποι οι οποίοι ε, κάνουν επιθέσεις στον κυβερνοχώρο και πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα ώστε να αυξηθεί η χνηλασιμότητα, η λογοδοσία, η ταχεία πρόσβαση για να είναι επιτυχημένες οι διώξεις. Διότι όσο οι εγκληματίες αυτοί θεωρούν ότι μπορούν και να αποφύγουν οποιαδήποτε κύρωση, δεν πρόκειται και να αποτραπούν διότι θεωρούν το κυβερνοέγκλημα μια επιλογή ελκυστική και εύκολη. Διεξάγεται συζήτηση λοιπόν και εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και με το ΝΑΤΟ για να ενισχυθεί η συνολική μας προσπάθεια αντιτρομοκρατιακού αγώνα. Φώτιγκα. Άκουσα για πρώτη φορά σχετικά με την κυβερνοαποτροπή κάποιες ιδέες από πολύ υψηλά ιστάμενα πρόσωπα αξιωματούχους του ΝΑΤΟ, ε, βρετανικής μάλιστα εθνικότητας. Ασφαλώς και πρέπει να συνεργαστούμε εν προκειμένου με το ΝΑΤΟ. Το οποίο είναι προχωρημένο στην προσπάθεια αυτή. Τάνοκ, είναι ενδιαφέρουσα η ιδέα αυτή κύριε Επίτροπε. Μπορείτε να επιβεβαιώσετε ότι όλες οι χώρες μέλη και οι πιο πρόσφατες ότι για όλες αυτές ε, ασχολούνται με το κυβερνοέγκλημα και την δίωξη. Γνωρίζω ότι η χώρα μας ασχολείται και υπάρχει ενδεχόμενο να γίνει μια, κάποια διεθνής διάσκεψη που να περιλάβει και χώρες όπως Κίνα Ρωσία σε βάση Ηνωμένων Εθνών. Αυτό ίσως είναι κάποια ρηξικέλευτες σκέψεις, αλλά γίνονται. Υπάρχει μια διεθνή σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης. Εμείς θα συνεχίσουμε να ζητάμε την ενίσχυσή της αν θέλετε, η ποινικοποίηση όλων αυτών των διαδικασιών, οι ποινικέ συνέπειε που μπορεί να υπάρξουν, οι κυρώσει κτλ. είναι θέματα τα οποία είναι υποσυζήτηση. Νομίζω ότι έτσι κλείσαμε τον κατάλογο των ομιλητών. Σας ευχαριστώ πολύ Επίτροπε για την ανταλλαγή των απόψεων. Ελπίζω να σας ξαναπούμε κατά τη διάρκεια της ε, περίοδου αυτής και σας ευχαριστώ και σας χειροκροτούμε.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 Έχουμε ακόμα ένα θέμα στην ημερήσια διάταξή μας, κυρίες και κύριοι. Ε, είχε ήδη αναβληθεί από την προηγούμενη συνεδρίαση. Είναι σημαντική διάσκεψη που οργανώνεται στο... Υπάρχει μάλλον ε, σημαντική διάσκεψη που οργανώνεται εδώ στο κτίριο του Κοινοβουλίου και γι' αυτό είναι πολύ άσχολοι οι συνάδελφοί μας. Ε, πρόκειται για αποστολή της ε, ΣΕΝΤΕ στην Ιαπωνία. Η επίσημη έκθεση είναι σχεδόν έτοιμη. Θα την διαβιβάσουμε, θα την διανύμουμε σχετικά σύντομα. Θα ήθελα τώρα να ολοκληρώσουμε το θέμα αυτό θυμίζοντας τα πιο σημαντικά γεγονότα σχετικά με την αποστολή αυτή που διεξήχθη τέλη Μαΐου, στο δεύτερο μισό του Μαΐου, με συμμετοχή πέντε ευρωβουλευτών από τις μεγαλύτερες πολιτικές ομάδες, μεταξύ αυτών και εγώ, η Ιδία, η κυρία Άννα Γκόμες, η κυρία Φρουζούλτσα από Σοσιαλιστές και Δημοκράτες, το Μπόγκταν επίσης, ο κύριος Ζέφρι Φαν Όρντεν από τους ε, συντηρητικούς, εγώ ίδια, πάλι από την ίδια πολιτική ομάδα και συνοδευθήκαμε από τον επικεφαλής της γραμματείας και ε, από ορισμένου ειδικού της γραμματείας και ένα αριθμό μεταφραστών. Πολύ υψηλού επίπεδου η αποστολή και πραγματικά έγινε ε, δεκτή με θαυμάσιο τρόπο από τους ε, Ιάπωνες αρμοδίους με επαφές με τον Υπουργό Εξωτερικών με άλλους αξιωματούχους του Υπουργείου Εξωτερικών, τον Υπουργό κ. Κίση, που είναι και αδελφός του Πρωθυπουργού και υπεύθυνο μεταξύ άλλων για ευρωπαϊκές υποθέσεις. Πρώτα συναντηθήκαμε με τον Υφυπουργό Άμυνας, σημαντικούς, ευρωβουλε... ε, σημαντικούς συγγνώμη, Ιάπωνες βουλευτές, μεταξύ αυτών και του επικεφαλής του Συνδέσμου Φιλίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι και υπουργό αρμόδιος για την ανάπτυξη, καθώς και με τον υπουργό Ισιχάρα και το Γενικό Γραμματέα του Συνδέσμου Φιλίας. Μας δέχθηκε και ο πρόεδρος της Επιτροπής Άμυνας της Ιαπωνικής Δίαιτας, καθώς και βεβαίως τέλος αλλού δόλος έσχατος, ένας αριθμός αξιωματούχων ε, της ε, Ιαπωνικής δύναμης αυτοάμυνας και ιδίως του ναυτικού, του Ιαπωνικού ναυτικού. Ε, μεταδίκαμε και, στο, και στην ναυτική σχολή, σχολή δηλαδή ναυτικών δοκίμων του Ιαπωνικού ναυτικού, που εκεί αποκαλείται ναυτική δύναμη αυτοάμυνας. Μεταβήκαμε και στην ναυτική βάση Ιωκοσούκα Επισκεφθήκαμε και ένα πολεμικό σκάφος στην ίδια αυτή βάση καθώς και το ναυπηγείο στην Ιωκοχάμα. όπου μπορέσαμε να παρακολουθήσουμε φάση κατασκευής πολεμικών σκαφών αλλά και μη στρατιωτικών, μη πολεμικών σκαφών. Ε, πολύ γενναιόδωρα μοιράστηκαν πληροφορίε μαζί μας οι κορεσπότες μας. Προβήκαμε και σε ανταλλαγή απόψεων με ανώτερους συμβούλους του Ιαπωνικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας και αξιολογήσαμε μαζί τους την κατάσταση ασφαλείας και στην νότια Κινέζικη θάλασσα αλλά και κατά μήκος ολόκληρης διαδρομής μέχρι, μέχρι την νότια Κινέζικη θάλασσα. Το καυτό θέμα που έθεσαν όλοι οι συνομιλητές μας είναι η κατάσταση ασφαλείας στην κορεατική Χερσόνησο και ιδίω οι επιθετικές πολιτικές του καθεστώτος της λαοκρατικής δημοκρατίας της Κορέας καθώς και οι απειλές η απειλή μάλλον που προέρχεται από, την, από τις κινέζικες απόπειρες εμπλοκής για τα νησιά Σενκάκου. Εκεί υπάρχουν αντιθέσεις που δεν έχουν ακόμη επιληθεί. Βεβαίως οι Ιάπωνες συνομιλητές μας ανησυχούν πολύ από τις εκτοξεύσεις πυράβλων και πυράβλων μάλιστα που εκτοξεύονται από σκάφη μέσα στην οικονομική ζώνη της Κινέζικης θάλασσας και βεβαίως ορισμένες από τις ανησυχίες αυτές ακούστηκαν και στη διάρκεια της ε, διασκέψης κορυφής G7. Και μάλιστα περιλήφθηκαν και στα τελικά συμπεράσματα. Στο έγγραφο που συντάχθηκε λοιπόν επιτόπου. Θεωρούμε πράγματι ότι η αξιολόγηση της κατάστασης ασφαλείας στη νότια και ανατολική κινέζικη θάλασσα είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο θα πρέπει να θέσουμε και στις επόμενες συναντήσεις της υποεπιτροπής μας. Υπάρχουν εξελίξεις, από όσο γνωρίζουμε, ορισμένα μέλη ενδιαφέρθηκαν πολύ για την δυνατότητα δημιουργίας συνασπισμών, συμμαχιών και για ασκήσεις που διεξάγονται στην περιοχή με συμμετοχή των Ιαπωνικών δυνάμεων. και άλλων χωρών. Έχουμε την πρόθεση να συνεχίσουμε τον διάλογο με τους Ιάπωνες. Η Ιαπωνία είναι διατεθειμένη να συνεχίσει τις αμυντικές προσπάθειες και να συμβάλλει σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θεωρούμε ότι είναι αξιολογότατη η συνεργασία αυτή και αναμένουμε να επιτεθεί πρόοδο στον διάλογο μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ιαπωνίας. Την επίσημη έκθεση της αποστολής θα σας την διαβιβάσουμε. Θεωρούμε ότι ήταν γενικώς επιτυχής η αποστολή αυτή και από τους Ιάπωνες οικοδεσπότες και από τη δική μας πλευρά. Ιδιαίτερος επιτυχής θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Γραμματεία της Υποεπιτροπής, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, ιδίως βεβαίω τον ε, πρέσβη στη επιτόπου, τους πρέσβεις και το προσωπικό τους στην Ιαπωνία για την υποστήριξή τους και βεβαίως είμαι ευγνώμων απέναντι στους Ιάπωνες οικοδεσπότες μας που υπήρξαν ιδιαίτερα γενναιόδοροι σε ό,τι αφορά την ε, συζήτηση μαζί μας των πληροφοριών. Θα ήθελα να κλείσω εδώ το θέμα αυτό. Δεν ξέρω αν οι ευρωβουλευτές επιθυμούν να συζητήσουν περαιτέρω το θέμα αυτό. Σας παρακαλώ πάντως, σας προσκαλώ να συμμετάσχετε στην αυριανή συνεδρίαση όπου έχουμε ορισμένα σημαντικά θέματα στην ημερήσια διάταξή μας και θα συνεχίσουμε με την έγκριση της εκθέσεως για τις εξαγωγές εξοπλισμών. Δεύτερη συζήτηση αυτή. Α, με συγχωρείτε, δεν σας είδα. Κύριε Κιούρεκ, ευχαριστώ αγαπητή Πρόεδρε. Ήρθα να σας ρωτήσω για την αποστολή που συζητήσατε. Μιλήσατε για ζητήματα ασφάλειας Τη Ταϊβάν. Ναι, συνομιλήσαμε για την Ταϊβάν με του Ιάπωνε. και εγώ μάλιστα μετέβη στην Ιαπωνία μετά από επίσκεψή μου στην Ταϊβάν όπου συναντήθηκα με τον Πρόεδρο, με τον Υπουργό Εξωτερικών και με πρώην Υπουργού Εξωτερικών. Άρα ήταν πολύ σημαντική η συζήτηση που διεξήχθηκε και στην Ιαπωνία για ζητήματα Ταϊβάν. Δεν έχω άλλες ερωτήσεις, ε, λέει η κυρία Φώτιγκα. Ας ολοκληρώσουμε λοιπόν την απογευματινή μας συνεδρίαση και σας προσκαλώ στην αυριανή συνεδρίαση που θα αρχίσει στις 9.30 το τελευταίο θέμα της ημερησίας διάταξης έχει ενδιαφέρον. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα συνάντηση με καναδική κοινοβουλευτική αντιπροσωπεία που επισκέπτεται την Ευρωπαϊκή Ένωση και ανταλλαγή απόψεων και με εκπροσώπους ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Σας ευχαριστώ και ευχαριστεί η Πρόεδρος και τους Γερμηνείς και οι Γερμηνείς ανταποδίδουν.